Good Καλώς ορίσατε, συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι. Καθίστε παρακαλώ. Έχουμε αφήσει να περάσει αρκετή ώρα και νομίζω μετά το ακαδημαϊκό τέταρτο μπορούμε να αρχίσουμε. Έχουμε εδώ μέλη της Επιτροπής μας και κυρίσω την έναρξη της σημερινής συνεδρίας της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης. Πρώτο θέμα, έγκριση της ημερήσιας διάταξης. Έχετε λάβει το σχέδιο της ημερήσιας διάταξης στους φακέλους σας και θα ήθελα να προσθέσω κάτι εδώ. Από τότε που σας απεστάλλει την περασμένη Δευτέρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 8 Ιουλίου έστειλε μια κατεξοδότηση πράξη προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η πράξη αυτή σας απεστάλλει επίσης στις 9 Ιουλίου με mail. Και πάλι ε, μας τριμώχνει κάπως ε, αυτό το χρονοδιάγραμμα γιατί βάσει των κανόνων που διέπουν τις κατεξουδότηση πράξης εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν αποφανθεί εντός δύο ημερολογιακών μηνών αυτή στιγμή διαβιβαστεί, άρα 8 Σεπτεμβρίου ή αν δεν ζητήσει παράταση της περίοδου αυτή, θεωρείται εγκεκριμένη εν λόγω πράξη. Γι' αυτό είμαστε υποχρεωμένοι να το εγγράψουμε σήμερα στην ημερήσια διάταξη. Και προτείνω να ασχοληθούμε ε, αύριο με αυτό το θέμα, να το εγγράψουμε ως τελευταίο θέμα στην ημερήσια διάταξη μετά την ανταλλαγή απόψεων που θα έχουμε με τον κύριο Κέσλερ. Συμφωνούμε? Ναι, ευχαριστώ πολύ. Άλλα σχόλια ή προτάσεις για την ημερήσια διάταξη έχουμε? Όχι. Ωραία. Άρα εγκρίνεται η ημερήσια διάταξη. Έγκριση των πρακτικών της συνεδρίασης 17 Ιουνίου 2015. Τα έχετε και αυτά στα χέρια σας, έχουν ε, διανεμηθεί και προτείνω ως συνήθω αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης να θεωρηθούν εγκεκριμένα τα πρακτικά. Σχόλια σχετικά έχουμε, όχι. Επόμενο θέμα. Ανακοινώσεις της Προέδρου. Έχω δύο ανακοινώσεις να σας κάνω και θα προσπαθήσω να είμαι πάρα πολύ σύντομη. Καταρχάς θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι σήμερα το πρωί συμμετείχα στη συνεδρίαση της Επιτροπής ΚΟΤΕΡ, της Επιτροπής Περιφερειών. Είχε την καλοσύνη να με προσκαλέσει για να κάνω μια παρουσίαση για το πώς λειτουργεί εδώ η Επιτροπή μας και με τι ασχολείται και να δούμε τι δυνατότητες υπάρχουν για καλύτερη συνεργασία και καλύτερο συντονισμό των δύο Επιτροπών μας. Χαίρομαι που όλα τα θέματα απασχολούν εμάς, απασχολούν και την Επιτροπή Κοτέρ τη Επιτροπής Περιφερειών, που είναι η ομόλογη Επιτροπή. Είχαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα ανταλλαγή απόψε και χαίρομαι για κάποιες ιδέες ε, που εκφράστηκαν για τη μελλοντική αγαστή συνεργασία των δύο Επιτροπών. Ανακοίνωση δεύτερη. Διάσκεψη των Προέδρων Επιτροπών συνεδρίασε την περασμένη εβδομάδα ενώ ήμασταν εμείς στο Στρασβούργο και κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης ανταλλάξαμε απόψεις με τον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον κύριο Τίμερμαν. Αυτό είναι πάγια συνεργασία που έχουμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να έχουμε στενότερη συνεργασία και ανταλλαγή απόψεων η διάσκεψη των Προέδρων των Επιτροπών με τον Αντιπρόεδρο Τίμερμαν. Κατά τη διάρκεια λοιπόν της συνεδρίασης εγώ έθεσα το ζήτημα των πολιτικών που βρίσκονται στο στάδιο της εφαρμογής και της υλοποίησης όπως είναι η πολιτική συνοχή και για τον καλό συντονισμό επίσης μίλησα μεταξύ των διαφόρων μέσων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ιδιαίτερα μια καλή συνεργασία μεταξύ των διαρθρωτικών ταμείων και του νέου Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων του Έχω τη χαρά να σας ε, πληροφορώ ότι ο κύριος Τίμερμαν συμφώνησε απολύτως. Είχαμε απόλυτη ταύτιση απόψεων και μας υποστηρίζει για την εφαρμογή της πολιτικής συνοχής. Επίσης ανέφερε ότι θα αποτελέσει και σημαντικό τμήμα του προγράμματος εργασίας Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2016. για να υπάρξει μια ανασκόπηση, μια επισκόπηση μάλλον, ε, του τρόπου με τον οποίο συνεργάζονται οι διάφορες αρμόδιες επιτροπές. Αυτά λοιπόν ενημερωτικά για το τι συνέβη τις περασμένες εβδομάδες και μέρες. Και τώρα θα συνεχίσουμε, περνάμε στο σημείο 4 στην ημερήσια διάταξη, η μερίδα σχετικά με την εδαφική διακυβέρνηση και πολιτική συνοχής. Θα ήθελα να σας θυμίσω ότι η Επιτροπή μας ζήτησε από την ε, ε, Υπηρεσία Μελετών που είναι το τμήμα 2, να ε, διοργανώσει ένα εργαστήριο για την εδαφική διακυβέρνηση. Είναι σχετικά νέα πολιτική αυτή και περιπλοκή και θα θέλαμε να την εξετάσουμε. Συνδυάζει δύο βασικά στοιχεία της πολιτικής συνοχής. Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση και τοπική προσέγγιση. Όπως βλέπετε και στο πρόγραμμα, σήμερα θα ακούσουμε τρεις παρουσιάσεις με διάφορα στοιχεία περιφερειακής διακυβέρνησης, εδαφικής, θα αρχίσουμε με μια εισαγωγή ε, της πολιτικής αυτής και πώς συνδέεται με την πολιτική συνοχής και την εφαρμογή της. Στη συνέχεια θα ακούσουμε για τις προοπτικές ε, της τοπικής αυτοδιοίκησης και τέλος θα δούμε ένα παράδειγμα ε, καλής πρακτικής επιτόπου όπως εφαρμόζεται στην περιφέρεια της Φλάνδρας. Έχουμε ως ομιλητές τον κύριο Κάι Μπέμε, και την κυρία Σουσάνε Τσίλμερ από το Ερευνητικό Κέντρο Special Foresight και τον κύριο Άμπελ Σούμαν από τον ΝΟΣΑ ε, για τη δημόσια δίκηση και την εδαφική ανάπτυξη και τον κύριο Ρενέ Φαντελέκ που είναι ο διαχειριστής του προγράμματος ε, στη συγκεκριμένη περίπτωση που θα εξετάσουμε για την περιφέρεια της Φλάνδρας. Μετά τις παρουσιάσεις θα δώσω το λόγο στα μέλη της Επιτροπής για σχόλια και ερωτήσεις. Προτείνω να αφιερώσουμε μια μισή ώρα ε, σε αυτή την ακρόαση και να ολοκληρώσουμε τις συζητήσεις μας στις 5 παρατέταρτο. Έχουμε λοιπόν εκπροσώπους και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής παρόντες από τη Γενική Διεύθυνση Ρέγγι. Είναι ο κύριος Μάρτον Ματκό. Δίνω λοιπόν αμέσως το λόγο στον κύριο Μπέμε και στην κυρία Τσίλμερ. Παρακαλώ. Good afternoon everybody. Σας ευχαριστώ και καλησπέρα σας. Η συνάδελφος Αμπίνε Τσίλμερ και ο υποφαινόμενος θα προσπαθήσουμε με μέσα στο τέταρτο που μας αναλογεί να σας κάνουμε μια σύντομη ανασκόπηση της εδαφικής διακυβέρνησης και το σχετισμό της με την πολιτική της συνοχής. Περίπλοκο θέμα, ελπίζω να σας ε, δώσουμε τροφή για σκέψη και να σας παρουσιάσουμε τις αδερές γραμμές ε, αυτού του θέματος. Δεν μπορούμε να επισέλθουμε να εντρυφήσουμε σε πολύ ε, λεπτομερή θέματα. Θα σας πούμε καταρχήν τι στη εδαφική διακυβέρνηση, πώς συνδέεται με την πολιτική συνοχής και ε, σε ποιο βαθμό μετά το πλαίσιο, τι μεταβλητές δημιουργεί και τι γίνεται με τις θεσμικές ικανότητες ό,τι αφορά την εδαφική διακυβέρνηση και πώς θα τις ενισχύσουμε. Θα ολοκληρώσουμε με τα ωφέλη και τις προκλήσεις Τη εδαφική διακυβέρνηση και πώ μπορούμε να την αναβαθμίσουμε, να την ενισχύσουμε. Ε, προς εξοικονόμηση χρόνου θα ξεκινήσω με το τι εστί εδαφική διακυβέρνηση και πώ μπορούμε να την ορίσουμε. Η Σαμπίνε θα προσπαθήσει να σα το εξηγήσει. Ήδη μα ε, είπατε αγαπητοί συνάδελφε ότι ε, η ότι δεν υπάρχει κάποιος ε, τέλειος ορισμός ε, ή οριστικός, ε, αλλά κάποιες βασικές έννοιες στις οποίες στηρίζεται η εδαφική διακυβέρνηση. Καταρχήν στηρίζεται στην πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, δηλαδή στην συνεργασία των διαφόρων φορέων της πολιτικής σε διάφορα επίπεδα διοικητικά και μια προσέγγιση που στηρίζεται στο τόπο, δηλαδή εστιάζεται στις ιδιαιτερότητες συγκεκριμένης εδαφικής επικράτειας. Και επίσης ε, έχει και πιο μακροπρόθεσμη στρατηγική προοπτική που δεν είναι μόνο κλαδική, μόνο τομεακή, αλλά λαμβάνει υπόψη και κοινωνικούς στόχους. Θα μπορούσαμε συνοψίζοντας να πούμε με απλά λόγια ότι η εδαφική διακυβέρνηση είναι μια χρηστή διακυβέρνηση που έχει σαφή σχετισμό και ενδιαφέρεται για τις ιδιαιτερότητες και τις ενισχύσεις συγκεκριμένου τόπου. Να δούμε όμως πώς συνδέεται η εδαφική διακυβέρνηση με την πολιτική συνοχής. Σας παραπέμπω στον συνάδελφο. Έχουμε καταρχήν μια ευρεία διασταλτική ερμηνεία της εδαφικής διακυβέρνησης και καλύπτουμε τις ε, τρεις διαστάσεις. Καταρχήν ε, την πρώτη που στηρίζεται στον τόπο, τη δεύτερη στη διακυβέρνηση και την τρίτη διάσταση που στηρίζεται στη στρατηγική πιο μακροπρόθεσμη προοπτική. Αυτές είναι οι τρεις διαστάσεις και επιλέξαμε και έξι στοιχεία της υφιστάμενης πολιτικής συνοχής. Και αφενός βλέπουμε τη θέσπιση ενός κοινού πλαισίου μια, ένα μεγαλύτερο προσανατολισμό προς τα αποτελέσματα για τη δεκαετία 2014-2020, μια θεματική συγκέντρωση, μια ενίσχυση της αρχής ε, της εταιρικότητας, εταιρικής σχέσης και επίσης η, ανάπτυξη των κοινοτήτων ε, στις, ε, και στις εδαφικές επενδύσεις, η, η διαχωρισμός της αστικής ανάπτυξης, της ανάπτυξης των πόλων, και επίσης ε, η μεταστροφή προ τα εθνικά προγράμματα σε σχέση με τα περιφερειακά. Αν αναλάβουμε λοιπόν αυτές τις έξι της ε, πολιτικής συνοχής και τις τρεις διαστάσεις που πιο αναλυτικά παραθέτονται και στο κείμενο, βλέπουμε ότι σε ό,τι αφορά την πρώτη διάσταση που στηρίζεται στον τόπο, ε, για την πρώτη περίοδο προγραμματισμού έχουμε ιδιαίτερη ενίσχυση της εταιρικής ε, σχέσης, της αρχής της εταιρικότητας και προσπαθούμε να δώσουμε μια πιο τοπική και περιφερειακή διάσταση σε αυτή την αρχή της εταιρικότητας. Σε ό,τι αφορά το CLLD και το ITI, σίγουρα και εδώ έχουμε τέτοια διάσταση ε, τοπική και για να είμαστε ειλικρινείς και ε, έντιμοι πρέπει να αναγνωρίσουμε τη, τη μικρή εμβέλεια αυτών των μηχανισμών, που είναι καλή, αλλά δεν έχουν επαναστατικά αποτελέσματα, πολύ περιορισμένα αποτελέσματα στην πολιτική συνοχή. Από την άλλη πλευρά, το 5% για την βιώσιμη ανάπτυξη πέθρου έχει στενή σχέση και με τα εδάφη στους συγκεκριμένους τόπους και η προσημείωση για τη αστική ανάπτυξη έχει μια ισχυρή διάσταση τοπική, αλλά σε ό,τι αφορά τη θεματική προσέγγιση έχουμε μεγάλες αφιβολίες ε, όπως έχει εφαρμοστεί για τα διαρθρωτικά ταμεία και το Ταμείο Συνοχής. Έχει περισσότερο ε, τομεακή διάσταση παρά τοπική διάσταση. Το ίδιο ισχύει και για την ε, μετατροπή, μεταστροφή προς τα εθνικά προγράμματα και τα περισσότερα κονδύλια που αφιερώνονται. Φυσικά υπάρχει ένα σχετισμό με του τοπικού και περιφερειακού εταίρου, αλλά όχι τόσο μεγάλο. Και σε ό,τι αφορά το κοινό πλαίσιο και την, τον προσανατολισμό στα αποτελέσματα, προ το παρόν είναι ουδέτερο προ την πρώτη διάσταση. Αυτά ω προ την πρώτη διάσταση. Τώρα, αν πάρουμε τη δεύτερη διάσταση τη ενίσχυση τη διακυβέρνηση και κυρίω τη πολυεπίπεδη και πολυτομεακή διακυβέρνηση, νομίζω ότι από αυτή την άποψη το κοινό πλαίσιο συνδυάζει διάφορα χρηματοδοτικά μέσα και έτσι ενισχύει την διακυβέρνηση και τη διάσταση διακυβέρνηση. Το ίδιο ισχύει για την αρχή τη Γιατί και εδώ φέρουμε κοντά διάφορους ε, ενδιαφερομένους και φορείς από πολλούς τομείς και τόπους, Το CLLD και τις ολοκληρωμένες εδαφικές επενδύσεις και εδώ έχουμε έμφαση το τοπικό σκέλος, πολύ χρήσιμο και σε ό,τι αφορά την προσημείωση, τον ειδικό προορισμό για τις πόλεις και αυτό ενισχύει τη διάσταση της διακυβέρνησης. Τώρα, για τη μεταστροφή στα εθνικά προγράμματα, νομίζουμε ότι ακριβώς επειδή αποδυναμώνεται το τοπικός και περιφερειακός ρόλος στην πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, δεν εξυπηρετεί την διάσταση της διακυβέρνησης. Το ίδιο και για τη θεματική συγκέντρωση. Αυτά σε αδρές γραμμές ε, τις λεπτομέρειες στο έγγραφό μας. Και τέλος, ε, τη στρατηγική για τη μακροπρόθεσμη διάσταση και πώς αυτή έχει ενισχυθεί. Εξετάσαμε όλους τους τομείς και θα μπορούσαν να ισχύουν προς τη μία ή την άλλη κατεύθυνση. Δηλαδή είτε να ενισχύουν είτε να αποδυναμώνουν αυτή τη διάσταση. ίσως ε, έχουμε καλύτερο προσανατολισμό, χρειαζόμαστε καλύτερο προσανατολισμό προς τα αποτελέσματα, κάτι που δεν εξυπηρετεί μέχρι στιγμής την ε, μακροπρόθεσμη στρατηγική διάσταση. Αλλά επαναλαμβάνω, ε, σε μεγάλο βαθμό όλα αυτά εξαρτώνται από τον τρόπο εφαρμογής, το, βαθμό εφαρμογής και το πώς θα διαχειρίζονται τα κράτη-μέλη τα διάφορα προγράμματα. Ε, στο πλαίσιο τώρα της εφαρμογής, ε, το πλαίσιο έχει ιδιαίτερη βαρύτητα. Και εκεί μπορούμε να ενισχύσουμε την εδαφική διακυβέρνηση και να αξιοποιήσουμε τις δυνατότητες. Και η συνάδελφος ε, θα σας πει για το ρόλο που έχει το πλαίσιο στην ενίσχυση της εδαφικής διακυβέρνησης. Φυσικά το πλαίσιο μετράει. Έχουμε διαφορετικά βέβαια είδη πλαισίου που μας ενδιαφέρουν εδώ. Καταρχήν το θεσμικό πλαίσιο, μιας χώρας, μιας περιφέρειας ε, ή μιας πόλης γιατί αυτό καθορίζει ποιος εμπλέκεται στην ε, διαδικασία της διακυβέρνησης, γιατί έχουμε διαφορετικό διαχωρισμό των ευθυνών ε, μεταξύ των τομέων και των περιφερειών και επίσης και ο ρόλος της κοινωνίας των πολιτών διαφέρει σε διάφορα μέρη της Ευρώπης. Δεύτερο πλαίσιο αφορά το, την παρακαταθήκη τις παραδόσεις, τις κυβερνητικές διαδικασίες. Ό,τι έχουμε κληρονομήσει λοιπόν, που επίσης είναι διαφορετικές. Και βλέπετε από τον πίνακα κάποιες ενδείξεις των διαφορών. Επίσης, οι δείκτες της Παγκόσμιας Τράπεζας ε, και η ειδική επισκόπηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, δείχνουν ε, ε, την πολιτική σταθερότητα, την αποτελεσματικότητα της πολιτικής, θέματα όπως η εμπιστοσύνη και βλέπουμε ότι είναι πιο θετική η κληρονομιά στις βορειότερες χώρες, ε, Σουηδία, Δανία και λιγότερο ευνοϊκές παραδόσεις σε τέτοιων διαδικασιών διακυβέρνησης ε, στην νότιο, σε μερικά τμήματα της Νοτιού Ευρώπης και στην Ανατολική Ευρώπη. Τρίτο πλαίσιο που μετράει είναι το κατά πόσο υπάρχουν μεμονωμένοι ε, εμπνευστές ε, άνθρωποι που προωθούν τέτοιου είδους διαδικασίες. Και τέλος, η παράδοση αφορά και τους τρόπους διακυβέρνησης. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι εφαρμογής των πολιτικών. Και μάλιστα εμείς διακρίνουμε μεταξύ τεσσάρων τρόπων που χρησιμοποιούνται σε διαφορετικό βαθμό και για διαφορετικές περιστάσεις και ανάλογα με το τι ε, γνωρίζουν οι φορείς, εφαρμόζουν και τους διαφορετικούς αυτούς τρόπους της διακυβέρνησης. Έχουμε τόσο διαφορετικά πλαίσια λοιπόν, που καθιστά δύνατη την ύπαρξη μιας ενιαίας λύσης ε, για όλους. Βέβαια, ίσως δεν είναι αυτή η πιο αρεστή πρόταση, αλλά θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τα διαφορετικά πλαίσια. Δεν έχουμε τόσο μεγάλες διαφορές τόσο διαφορετικά πλαίσια, διαρωτόμαστε τι είδου ε, θεσμικέ ικανότητε χρειαζόμαστε. Σε ό,τι αφορά θεσμική ικανότητα, θεσμικές ικανότητες, ε, θα πρέπει να έχουμε υπόψη ότι δεν είναι πανάκια οι γρήγορε οι τη της διακυβέρνηση. Είναι χρονοβόρε και απαιτούν και πόρου και χρόνο για να εξασφαλίσουμε ενεργό συμμετοχή πολλών φορέων. Και σε ό,τι αφορά τη θεσμική ικανότητα, έχουμε δύο είδη φορέων. Καταρχήν χρειαζόμαστε μια υπεύθυνη ηγεσία. Και είναι σημαντικό να υπάρχει σαφή διάκριση των ρόλων και των ευθυνών. Για να ξέρουν οι φορεί πώς λειτουργεί το σύστημα και να μπορούν να το χρησιμοποιούν. Και το θέμα και της ε, ανάληψης τη εξουσίας, χειραφέτησης ε, της ηγεσία. Θα πρέπει και οι μεμονωμένοι ε, ιδιώτες και οι θεσμοί να έχουν την εξουσία να εφαρμόσουν αυτές τις πολιτικές. Και επίσης θα πρέπει να δούμε να, πώς θα αναγνωρίσουμε τέτοιους ικανούς φορείς. Είναι σαφές ε, στη διαδικασία ποιος αναλαμβάνει τον ηγετικό ρόλο και ποιος την προωθεί. Επαναλαμβάνω, μπορεί να είναι ιδιώτη αυτός ε, ή θεσμό. Θα πρέπει όμω να έχει ικανότητε για να αναλάβει τον ηγετικό ρόλο. Ιδιαίτερα στην μακρόχρονη περίοδο που χρειάζεται για τη διακυβέρνηση. Ε, δεν μας ε, ενδιαφέρει μόνο η ηγεσία όμως, αλλά και η συμμετοχή. Γιατί έχουμε συνήθως πολλού φορεί που χρειάζονται και χρόνο και πόρους και ικανότητες ε, νοητικές ε, για να συμμετέχουν στη διαδικασία. Μερικές φορές λείπουν αυτά τα στοιχεία. Επίσης, ε, σε ό,τι αφορά τη θεσμική ικανότητα των ενδιαφερομένων φορέων θα πρέπει να υπάρχει στην ελαφρική διακυβέρνηση. Είναι σημαντικό αυτό το στοιχείο. Ορίζουμε ότι υπάρχουν κάποιες αλλαγές. Χρειαζόμαστε κάποια ευελιξία αλλά ταυτόχρονα και ασφάλεια δικαίου. Γιατί μπορεί να αλλάζουν και οι φορείς, οι ρόλοι του ίδιου φορέα, αλλά παρά την ευελιξία που είναι απαραίτητη, χρειαζόμαστε ταυτόχρονα και μια ασφάλεια δικαίου. Γνωστές και ασφαλείς συνθήκες ε, για το νομικό πλαίσιο, για το δικαιωτικό πλαίσιο. Και επίσης ε, να εστιαστούμε στην ε, θεσμική προσαρμοστικότητα να ξέρουμε ότι οι θεσμοί μπορούν να προσαρμόζονται στη διαδικασία και να προβούν στις απαραίτητες αλλαγές. Οπότε η θεσμική ικανότητα είναι σημαντικό θέμα και απαιτεί και τους απαραίτητους πόρους. Οπότε πριν ξεκινήσουμε τη διαδικασία της εδαφικής διακυβέρνησης θα πρέπει να γνωρίζουμε σαφήνεια γιατί το κάνουμε, ποια είναι τα ωφέλη αυτής της εδαφικής διακυβέρνησης, ποιες είναι οι προκλήσεις και θα μας εξηγήσει το περαιτέρω η Σαμπίνε. Όπως είπα στην αρχή, ένα χαρακτηριστικό του συστήματος εδαφικής διακυβέρνησης είναι ότι έχει μία μακροπρόθεσμη στρατηγική στρατηγική που εξυπηρετεί τους κοινωνικούς στόχους. Αυτό σημαίνει ότι δεν είναι στόχος η ίδια, αλλά είναι ένα μέσο για την επίτευξη άλλων στόχων. Ακολουθώντα μια τέτοια προσέγγιση, είμαστε σε θέση να λάβουμε καλύτερη υπόψη τις εδαφικές ιδιαιτερότητε. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ε, το εδαφικό δυναμικό καλύτερα και να γνωρίζουμε πού ε, έγκυζε τα προβλήματα. Και Μπλέκοντας όλους τους αρμόδιους για τη λήψη αποφάσεων μπορούμε να ενσωματώσουμε διάφορες πολιτικές και να, δι... και να τους ε, κάνουμε να ιδιοποιηθούν αυτές τις ε, πολιτικές γιατί συμμετέχουν και ταυτόχρονα να αναγνωρίσουμε διάφορους στόχους διαφορετικών τομέων, διαφορετικών επιπέδων. Οι φορείς λοιπόν το συνειδητοποιούν αυτό και αργά ή γρήγορα θα πρέπει να δραστηριοποιηθούν και να μην κλείνουν πια τα μάτια τους και να αρνούνται την κατάσταση. Όπως είπε ο Κάι ήδη, ταυτόχρονα είναι πολύ ε, ενδιαφέρον, είναι χρονοβόρο, απαιτητικό όσον αφορά ε, το δυναμικό και οδηγεί σε μια μεγάλη ποικιλία διαφορετικών προσεγγίσεων για διαφορετικά μέρη και διαφορετικές πολιτικές. Και έτσι φτάνουμε στο ερώτημα τι μπορούμε να κάνουμε ώστε να ξεπεράσουμε αυτές τις προκλήσεις και να ενισχύσουμε την εδαφική ε, διακυβέρνηση εφόσον ε, βοηθά στην επίτευξη των γενικών μας στόχων. Κλείνοντας, θα πρέπει να θυμίσουμε ότι η εδαφική διακυβέρνηση δεν είναι αυτός σκοπός. Πρέπει να ξεκινήσουμε από την ανάγκη ότι υπάρχουν διάφορα επίπεδα προβλημάτων που πρέπει να επιληθούν και με την με την εδαφική διακυβέρνηση μπορούμε να έχουμε πιο αποτελεσματικές και αποδοτικές λύσεις από ότι οι ε, στάνταρ διαδικασίες. Το βασικό είναι ότι δεν είναι αυτός ο σκοπός είναι η εδαφική διακυβέρνηση μπορεί να είναι η καλύτερη κατάλληλη προσέγγιση. Και έπειτα εξετάζοντας διάφορα παραδείγματα στην Ευρώπη και έχουμε κάποια και στο εγγραφό μας, Βλέπουμε πως εν τέλει χρειάζεται μια νέα νοοτροπία στο δημόσιο τομέα, μετακίνηση από την απόδοση που έχει προσανατολισμό τη συμμόρφωση σε μια ε, ε, απόδοση που έχει στόχο τα αποτελέσματα. Δηλαδή πιο πολύ επιχειρηματικό πνεύμα χρειάζεται. Μια τέτοια ε, νοοτροπία χρειάζεται. Αναφέραμε επίσης ότι θα πρέπει να χειραφετηθούν οι άνθρωποι που μπορούν να συγκεντρώσουν τους ενδιαφερόμενους φορείς, που μπορούν να έχουν ε, ε, την ε, στήριξη για να το καταφέρουν αυτό. Και τέλος, σε μια μελέτη που δημοσιεύθηκε πέρυσι από την ΕΣΠΟΛ, καλύπτουμε την εικόνα αυτή εξετάζουμε το πώς μπορούμε να υπερασπίσουμε και να στηρίξουμε την περιφερειακή, την εδαφική διακυβέρνηση με τέσσερις άξονες, συντονίζοντας δηλαδή τις δράσεις των φορέων και των θεσμών, ε, ολοκληρώνοντας τις διάφορους τομείς της πολιτικής, κινητοποιώντας τη συμμετοχή των βλεκομένων ε, φορέων και να μπορούμε να προσαρμοστούμε σε μεταβαλλόμενα πλαίσια. Δηλαδή δεν είναι πάντα η κατάλληλη ομοιόμορφη προσέγγιση και πρέπει να μπορούμε να προσαρμοστούμε, να υπάρχει δηλαδή ένας βαθμός ευελιξίας. Και επίσης διαρκώς να σκεφτόμαστε τον αντίκτυπο σε κάθε συγκεκριμένο χώρο των πολιτικών που προωθούμε. Πέντε σημεία κλειδιά λοιπόν που μας οδηγούν στο να προχωρήσουμε προς περισσότερη εδαφική διακυβέρνηση. Αυτά λοιπόν πολύ σύντομα, ε, γιατί είχαμε μόνο 15 λεπτά και προσπαθήσαμε να σας δώσουμε κάποια βασικά στοιχεία σε μια περίπλοκη. Είναι σαν διαφημιστικό για έναν έργο. Ελπίζω έτσι να λειτουργήσει και για σας και να κινητοποιήσει τη συζήτηση. Ευχαριστώ. Ναι, σχεδόν 15 λεπτά. Ναι, όντως πρόκειται για ενδιαφέρουσα βάση για συζήτηση. Τώρα θα συνεχίσουμε. με τον κύριο Σούμαν. με την παρουσίασή σας για την πολυπίπεδη, τα πολυ, συστήματα πολυπίπεδης διακυβέρνησης και τις μεταρρυθμίσεις στις τοπικές κυβερνήσεις. Μάλιστα. Καταρχήν σας ευχαριστώ που με καλέσατε σε αυτό το εργαστήριο για να σας παρουσιάσω την εμπειρία του ΟΣΑ και ίσως το πιο σημαντικό να πούμε εξ αρχή είναι ότι ο ΣΑ έχει ευρύτερη συμμετοχή από ότι οι, τα, οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οπότε παρουσιάζω αριθμούς και στατιστικές, δεν αφορούν μόνο την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά όλα τα κράτη του ΟΣΑ που περιλαμβάνουν και χώρες της Βόρειας Αμερικής, την Αυστραλία, το Ισραήλ, ε, τη Χιλή και χώρες της Ανατολικής Ασίας. Αν δούμε λοιπόν την υποεθνική, τις υποεθνικές κυβερνήσεις, ε, το πρώτο που έρχεται στο μυαλό μας είναι ότι έχουμε τεράστιο αριθμό υποεθνικών κυβερνήσεων. Σε ολόκληρο τον όσα έχουμε σχεδόν 140.000 μεμονωμένες ε, υπό εθνικές κυβερνήσεις. Δύο χώρε είναι αυτέ που ξεχωρίζουν ιδιαίτερα. Από τη μια πλευρά έχουμε τι ΗΠΑ και από την άλλη έχουμε τη Γαλλία, όπου έχουν περίπου 40.000 υπό εθνικές κυβερνήσεις αυτές οι δύο χώρε. κάθε μια από αυτέ τι δύο χώρε. Στην ΣΥΠΑ είναι μεγάλη χώρα βέβαια με 320, 320 εκατομμύρια κατοίκους ενώ στην Γαλλία έχουμε ένα τεράστιο αριθμό δήμων. Πάνω από το 1 τέταρτο των Δήμων από το σύνολο των Δήμων στον Οσάνικο στη Γαλλία. Έχουμε λοιπόν 135.000 δημοτικές αρχές στον ΟΣΑ, 5.000 περιφέρειες, ε, συγγνώμη, 500 περιφέρειες και 4.000 ενδιάμεσα επίπεδα τοπικών ε, κυβερνήσεων, που είναι κάπου ανάμεσα στο περιφερειακό και στο τοπικό επίπεδο διακυβέρνησης. Όταν τώρα εξετάσουμε λίγο πιο λεπτομερώς πώς ε, προσεγγίζουν τις υποεθνικές κυβερνήσεις στα διάφορα κράτη, ε, έχουμε χώρες σε δύο διαστάσεις. Καταρχήν έχουμε τη γνωστή ε, διάκριση ανάμεσα στις ομοσπονδίες <clears throat> και τις ενοποιημένες χώρες και μετά γίνεται και μία διάκριση ανάλογα με τα διάφορα υποεπίπεδα υποεθνικής ε, κυβέρνησης. Έχουμε χώρες όπου έχουν ένα επίπεδο υπό εθνικής διακυβέρνησης που είναι συνήθως οι Δήμοι. Έχουμε χώρες με δύο επίπεδα όπου υπάρχουν δηλαδή περιφέρειες ή κρατήδια και μετά τις, ε, τους Δήμους και μετά έχουμε και λίγες χώρες όπου υπάρχουν τρία διαφορετικά επίπεδα υποεθνικής κυβέρνησης. Έχουμε δηλαδή την περιφέρεια, το κράτος, κάποιο διάμεσο επίπεδο και μετά τους Δήμους. Όταν εξετάζουμε αυτές τις διάφορες χώρες λοιπόν υπάρχει μια σαφή στάση. Όσο μεγαλύτερη είναι η χώρα τόσο περισσότερα επίπεδα υποεθνικής ε, κυβέρνησης υπάρχουν. Αυτό είναι λογικό και αντικατοπτρίζει τα όσα είπαν οι προηγούμενοι ομιλητές, ότι δηλαδή δεν είναι δυνατόν να έχουμε μία ομοιόμορφη προσέγγιση για όλες τις χώρες και να εντοπίσουμε ποιο είναι το καλύτερο σύστημα υπεθνική διακυβέρνησης, αλλά ότι πρέπει πραγματικά να δούμε την εικόνα της κάθε χώρας και να βρούμε και το κατάλληλο σύστημα υποεθνικής διακυβέρνησης. Θα πρέπει επίση να εξετάσουμε ποιο είναι το πρώτο επίπεδο εθνική διακυβέρνηση, δηλαδή η περιφέρεια ή το κρατήδιο. Σε αυτό το γράφημα βλέπουμε το μέσο γεωγραφικό μέγεθος και το μέσο πληθυσμιακό μέγεθος μιας των, των διαφόρων χωρών του ΩΣΑ και υπάρχουν τεράστιες διακοιμάνσεις και διαφοροποίησεις. Έχουμε χώρες όπως η Ελβετία, η Ουγγαρία, η Τεχία, όπου η κάθε περιφέρεια είναι λίγα τετραγωνικά χιλιόμετρα, με λίγες χιλιάδες κατοίκους και μετά έχουμε χώρες, πολλές, που δεν υπάρχουν καν σε αυτό το γράφημα, διότι βρίσκονται τόσο απομακρυσμένες, είπα, όπου ε, μια πολιτεία έχει διάφορες εκατοντάδες χιλιάδες ε, τετραγωνικά μέτρα και κάποια εκατομμύρια κατοίκους. Το ίδιο και για τη Γερμανία, όπου το χαρακτηριστικό επίπεδο υποεθνικής κυβέρνησης ε, περιλαμβάνει 5 εκατομμύρια κατοίκους. δεν μας ενδιαφέρει μόνο η, κατανομή των χωρών σε υποεθνικές κυβερνήσεις, αλλά μας ενδιαφέρει και πόση εξουσία έχουν στη κατοχή τους. Και αυτό μπορούμε να το κρίνουμε από τις δημόσιες δαπάνες στις οποίες προβαίνουν αυτά τα διάφορα επίπεδα διακυβέρνησης. Αυτό που βλέπουμε στο φωτογράφημα είναι οι δαπάνες των υποεθνικών κυβερνήσεων σε σχέση με το σύνολο του ΑΕΠΑ. Και εδώ υπάρχουν τεράστιες ε, διακοιμάσεις. Στη Δανία, ας πούμε, το 60% των δημοσίων δαπανών γίνεται από τις εθνικές κυβερνήσεις, ενώ χώρες όπως η Ελλάδα, η Χιλή, η Νέα Ζηλανδία, μόνο γύρω στο 10% των δημοσίων δαπανών γίνεται από τις υποεθνικές κυβερνήσεις. Σχόλιο εκτός μικροφώνου. Um, βεβαίω, ε, εδώ έχουμε ένα τρόπο, ένα είδο μέτρησης εξουσίες και ευθυνών που φέρουν οι υποεθνικέ κυβερνήσεις, αλλά βεβαίω το γράφημα αυτό δεν μας λέει όλα τα στοιχεία γιατί είναι σημαντικό να ξέρουμε πώς θα δαπανούν οι κυβερνήσεις, αλλά και πόση αυτονομία έχουν στο να αποφασίσουν πώς θα τα δαπανήσουν όλα αυτά. Σε αυτό το γράφημα λοιπόν βλέπουμε ότι στις βόρειες σκανδιναβικές χώρες, Δανία, Σουηδία, Φιλανδία, έχουν ένα τεράστιο μερίδιο των δαπανών οι υποεθνικές κυβερνήσεις, όμως έχουν σχετικά μικρή αυτονομία. Γιατί έχουν πολύ ξεκάθαρα ε, καθήκοντα και λειτουργίες που πρέπει να εκπληρώσουν. Δαπανούν λοιπόν αυτά τα χρήματα που είναι πολλά, αλλά ε, δεν αποφασίζουν αυτές. Σας μίλησα λοιπόν περισσότερο για τις περιφέρειες και τα κράτη και τώρα θα ήθελα να μιλήσω για το δημοτικό επίπεδο. Και εδώ θα ήθελα να εστιάσω κυρίως στις αστικές, μεγάλες αστικές περιοχές και θα ήθελα να εστιάσω σε αυτές διότι οι ε, μεγάλες αστικές περιοχές, οι Μητροπόλεις είναι πολύ ιδιαίτερες. Και είναι πολύ σημαντικό το πώς δομείται η, τοπική κυβέρνηση, ο Δήμος. Εδώ έχουμε περιοχές που είναι πολύ στενά συνδεδεμένες όσον αφορά τις λειτουργικές διασυνδέσεις και τις κοινωνικο-οικονομικές διασυνδέσεις. Όλοι όσοι ζούμε σε μεγάλα αστικά κέντρα γνωρίζουμε πολύ καλά ότι ε, ζούμε σε ένα μέρος, ε, ε, εργαζόμαστε σε ένα άλλο, πάμε για ψώνια σε ένα παράλλο και ακόμα και επισκεφτόμαστε φίλους μας σε άλλο. Ε, το ίδιο και για τις επιχειρήσεις ισχύει που λειτουργούν σε ολόκληρη την αστική περιοχή. Αυτό που είναι αλήθεια όμως είναι για ολόκληρο τον ΩΣΑ είναι ότι αυτές οι λειτουργικές σχέσεις σχεδόν ποτέ δεν αντικατοπτρίζονται στο, στη θεσμική δομή των αστικών κέντρων. Συνήθως αποτελούνται από ανεξάρτητους δήμους. Και αυτό που βλέπουμε σε αυτό το γράφημα είναι ο αριθμός των Δήμων ανά 100.000 κατοίκους. Αν σκεφτούμε κάποιο αστικό κέντρο με 100.000 κατοίκους ας πούμε, θα δούμε ότι υπάρχουν πολλές μεγάλες αστικές περιοχές σε ολόκληρο τον ΩΣΑ και φυσικά στην Ένωση, όπου υπάρχουν δεκάδες ή και εκατοντάδες δήμοι. Και αυτό προκαλεί προβλήματα. Γιατί κάποιε από τις πολιτικές πρέπει να συντονίζονται ανάμεσα στου διάφορους δήμους. Για παράδειγμα, οι μεταφορές πρέπει να συντονίζονται. Επίση η χρήση των γεών, Δημόσιε υπηρεσίες πρέπει να συντονίζονται αν, θέλουμε να είναι αποτελεσματικέ και οικονομικές. Όταν έχουμε λοιπόν δεκάδες ή και εκατοντάδες δήμους, αυτό δημιουργεί τριβές και προκλήσεις. Αυτές οι τριβές που οφείλονται στο γεγονός ότι οι διοικητικές δομές δεν, δεν αντιστοιχούν στις λειτουργικές δομές, οδηγούν σε πολλές μεταρρυθμίσεις όπως αυτές που είδαμε τα τελευταία χρόνια και ιδιαίτερα στο επίπεδο των αστικών κέντρων. Υπήρξε μια τεράστια τάση σε, σε όλες τις χώρες του να γίνουν μεταρρυθμίσεις διακυβέρνησης ώστε να δημιουργηθεί ένα σύστημα διακυβέρνησης το οποίο να αντικατοπτρίζει καλύτερα αυτή την ε, λειτουργική αλληλεξάρτηση που παρατηρείται στα μεγάλα αστικά κέντρα. Ας πούμε σε χώρες που ε, προέβησαν στο πιο ριζοσπαστικό βήμα, δηλαδή τη συγχώνευση διαφόρων δήμων, αλλά παρατηρήσαμε συχνά ότι υπήρξαν και προσεγγίσεις για να δημιουργηθούν αρχές κάθε φορά στα αστικά κέντρα που είναι πάνω από το επίπεδο του Δήμου και που στόχο έχουν ακριβώς να συντονίζουν τις πολιτικές των διαφόρων δήμων μεταξύ τους. Αυτή η προσέγγιση ήταν αρκετά επιτυχής. Και έχουμε πράγματι στοιχεία στη διάθεσή μας που δείχνουν την επιτυχία αυτή. Και ίσως αυτό να είναι και το πιο, κοντά, πιο, πιο κοντινό, η πιο κοντινή προσέγγιση στην ομοιομορφία που λέγαμε. Δηλαδή καλύτερη, ε, ε, καλύτερο συνδυασμό του διοικητικού πλαισίου με το πραγματικό λειτουργικό πλαίσιο. Τα αποτελέσματα δηλαδή εδώ και 15-20 χρόνια είναι πολλά υποσχόμενα. Αυτά λοιπόν από μένα. Έχουμε και κάποιες άλλες δημοσίευσεις για τα ζητήματα αυτά αν σας ενδιαφέρουν και φυσικά με τα χαρά είμαι στη διαθεσή σας να απαντήσω ερωτήσεις. Ευχαριστώ. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ και τώρα συνεχίζουμε με τη Φλάνδρα και τον κύριο Ρενέ Βαντεβλέκ για την εδαφική διακυβέρνηση στην περιφέρεια της Φλάνδρας. Έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ που με καλέσατε. Είναι πολύ μεγάλη ευκαιρία που έχω να συνδέσουμε την Ευρωπαϊκή Πολιτική Συνοχής και τις περιφερειακές ε, πρακτικές, διότι είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό για να είναι οι πολιτικές πιο αποτελεσματικές σε όλα τα επίπεδα. Αρχίζω με μερικά βασικά στοιχεία ενημερωτικά για το σχέδιο μας το ρυθμιστικό του, του βορείου ε, άκρου των Βρυξελών. Έχουμε ένα νέο σχέδιο χωροταξικό. Ε, καταλήξαμε ότι πολλές από τις νέες ιδέες πρέπει να δοκιμαστούν και τις προσεγγίξεις για τη χάραξη πολιτικής. Και χρειαζόμαστε κάπου αυτό να το δοκιμάσουμε, να κάνουμε ένα τεστ. Και είπαμε ας χρησιμοποιήσουμε ε, ένα από τα εδάφη μας που έχουν ε, την περισσότερη κίνηση και τη μεγαλύτερη περιπλοκότητα που είναι αυτό το βόρειο ε, άκρο των Βρυξελών. Το όριο. Ε, η προετοιμασία άρχισε από το 2012, αλλά χρειάστηκε ε, λίγος καιρός για να ξεκινήσει το πρόγραμμα τον Αύγουστο του 2013 επίσημα. Για να ε, ρυθμίσουμε όλα τα ζητήματα. Και ξεκίνησε τότε επίσημα, δηλαδή εγκρίθηκε ο επικεφαλής και η ομάδα που θα λειτουργούσε, όπως επίσης και ο προϋπολογισμός του προγράμματος. Αυτό που έχει πολύ μεγάλη σημασία ε, είναι ε, να ξέρουμε ότι ε, είναι παραμεθόρια αυτή η περιοχή, συνορεύει με την περιφέρεια των Βρυξελών και χρειάστηκε να κάνουμε μια συμφωνία με την περιφέρεια των Βρυξελών και την επαρχία του φλαμαντικού Μπραμπάντ. Είχαμε ε, συγκεκριμένα στοιχεία και στόχους, πάρα πολύ βασικούς αλλά και πάρα πολύ σημαντικούς. Ένας από τους στόχους είναι να έχουμε ένα όραμα κοινό, μακροχρόνιο για την ανάπτυξη της περιφέρειας, αλλά είπαμε να μην περιμένουμε να βρούμε το όραμα πριν αρχίσουμε να ενεργούμε και να δραστηριοποιούμεθα. Δηλαδή, ε, υπήρχαν ήδη πολλά έργα σε αυτή τη γεωγραφική περιοχή, ε, σε αυτό το, το σύνορο Φλάνδρας και Βρυξελών και θελήσαμε να ε, συνδέσουμε και τα προγράμματα μεταξύ τους, τα έργα που ήδη έτρεχαν. Για χρησιμοποιείται ε, η περιφερειακή ανάπτυξη ως μοχλός γενικότερης ανάπτυξης και θα σας πω πώς αυτό λειτουργήσε. Προχωρούμε στην επόμενη διαφάνεια. Να δούμε λίγο το περιεχόμενο του έργου αυτού και του σχεδίου μας. Ποιο ήταν το πρώτο βήμα λοιπόν. Προσπαθήσαμε να καθορίσουμε ε, στόχους ε, με βάση τις τοπικές ανάγκες, αρχίζοντας από κάποιους γενικότερους στόχους ε, και μετά ένα ειδικό ρυθμιστικό αναπτυξιακό σχέδιο. Γενικοί στόχοι λοιπόν συζητήθηκαν σε ομάδες ενδιαφερομένων ε, για να μεταφραστούν επί τόπου κάθε φορά στην πράξη με προτεραιότητες και ιεράρχηση αυτών. Για ε, το ε, βόρειο σύνορο λοιπόν των Βρυξελών θέλαμε να αναζωογονηθεί δημογραφικά η περιοχή γιατί συχνά ήταν εγκαταλελειμμένη. μείωση της χρήσης επίσης των φυσικών πόρων, ιδιαίτερα των γεών γιατί έχουμε πρόβλημα έλλειψης γεών στην περιοχή. Και επίσης θέλαμε να βελτιώσουμε ε, τις συνθήκες διαβίωσης στο περιθώριο εκεί, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά ε, την υγεία ε, του πληθυσμού. Ε, είναι ο δακτύλιος εκεί αυτοκινητοδρόμου των Βρυξελών με πάρα πολύ μεγάλη κίνηση και ε, προβλήματα. Ε, θελήσαμε να αυξήσουμε την κοινωνική συνοχή και την ε, λειτουργική συνοχή και νέες οικονομικές δραστηριότητες να φέρουμε πιο μακροπρόθεσμα πάντα για την περιφέρειά μας. Of course, it's not... Βεβαίως. Εδώ βλέπετε στη διαφάνεια ε, την περιοχή αυτή που είναι ε, η το σύνορο Φλάνδρας Βρυξελών ε, προς το βοράν. Αναπτύξαμε κάποιες αρχές για την χωροταξία μας και το σχεδιασμό μας. Για να υπάρχει ένα κοινό όραμα, όπως είπαμε και προηγουμένως, αλλά θα πρέπει εκτός από οράματα να επιφέρουμε και αλλαγές και να κάνουμε στην πράξη κάποια ε, επιτεύγματα. Πώς γίνεται αυτό τώρα. Έχουμε μακρά προϊστορία ε, με την επικουρικότητα, αλλά πέρα από την επικουρικότητα συναντήσαμε στην πράξη ότι δεν λειτουργεί πια με την παλιά έννοια επικουρικότητα. Σήμερα έχουμε πολυεπίπεδη διακυβέρνηση και οι κυβερνήσεις συνεργάζονται ε, με επιχειρήσεις, ιστιτούτα, ιδιώτες, δίκτυα δημιουργούν, δεν είναι ανεξάρτητοι δεν είναι ελεύθερα ηλεκτρόνια. Είναι πολύ περίπλοκη η ανάπτυξη ενός ε, ε, εδάφους μιας επικράτειας. Δεν είναι απλή διακυβέρνηση. Θα πρέπει λοιπόν να δεχθούμε και να μάθουμε ότι υπάρχουν διαφορές απόψεων, δεν συμφωνούν όλοι σε μια επικράτεια και ε, πέρα από το κοινό όραμα χρειάζεται και διαπραγμάτευση για να αναπτύξουμε την περιοχή μας. Δηλαδή Υπάρχει το ύψιστο ε, αγαθό ε, που είναι το κοινό συμφέρον και πάντα θα πρέπει να αναζητούμε συνενέσεις και συμβιβασμούς. Δεν έχει δίκιο ένας κάθε φορά. Ούτε θα πρέπει ένας που αντιτίθεται σε ένα έργο να μπορεί να το μπλοκάρει στο σύνολό του. Αυτό ε, ε, μπορεί να είναι και κυβέρνηση, υψηλότερο ή χαμηλότερο επίπεδο διακυβέρνησης που αντιτίθεται. Οπότε δεν θα πρέπει το υψηλότερο επίπεδο διακυβέρνησης να είναι εκείνο που μπλοκάρει. Ε, βλέπουμε λοιπόν τα σύνορα Φλάνδρας Βρυξελών. Έχουμε εκεί 70 έργα παρακαλώ με 30 διαφορετικούς εμπνευστέ και φορείς και συμμετέχουν πάρα πολλά επίπεδα διακυβέρνησης ε, που είναι το, η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά το αεροδρόμιο, δύο αυτόνομες περιφέρειες που συνορεύουν εκεί και αυτό περιπλέκει τα πράγματα ε, γιατί έχουν ανταγωνισμό μεταξύ τους, έχουν διαφορετική κουλτούρα και ιστορία και όπως ξέρετε έχουμε και γλωσσικές εντάσεις στη δική μας περίπτωση. Επίσης υπάρχει μία ε, επαρχία και γύρω στους 20 δήμους. Καταλαβαίνετε πόσα επίπεδα διακυβέρνησης και βέβαια τα εδάφη της επικράτειας δεν τις φτιάχνουν οι θεσμοί, οι κυβερνήσεις, αλλά ο κοινωνικός ιστός, οι επιχειρήσεις, οι πολίτες, Ινστιτούτα, πανεπιστήμια, διάφορα συμφέροντα που θα πρέπει όλα αυτά να συγκεραστούν. Έτσι, ε, από εκεί ξεκίνησε και ήταν βασική ιδέα του προγράμματος. Τι κάναμε λοιπόν. Εκπονήσαμε μια στρατηγική ε, σε τρεις γραμμές δράσης. Πρώτον, συνεργασία, σας το είπα ήδη, αρχίσαμε από αυτή τη βασική συμφωνία σε διασυνοριακό επίπεδο με την περιφέρεια των Βρυξελών, εμείς η περιφέρεια της Φλάνδρας και στην αρχή καλέσαμε όλους τους ενδιαφερομένους που είναι πολλοί και δραστηριοποιούνται εκεί για να δημιουργήσουμε μια πλατφόρμα και να βεβαιωθούμε ότι λαμβάνονται υπόψη όλα τα συμφέροντα και ε, μπορούν να συνεργάζονται οι ενδιαφερομένοι σε ομάδες εργασίας κτλ. Το δεύτερο επίπεδο ήταν ε, ή σε μια δεύτερη φάση ε, κάναμε έρευνα, ε, συλλέξαμε ιδέες και τα φέραμε αντιμέτωπα με την πραγματικότητα κάθε φορά. Και ε, καταφέραμε έτσι με πραγματική χαρτογράφηση να φωτογραφίσουμε την κατάσταση και να δούμε πώς μπορούμε να συνδέσουμε έργα διαφόρων ε, φορέων να αποκτήσουν έτσι μια εικόνα, οπτική απεικόνηση, χαρτογράφηση για να καταλάβει ο κόσμος περί πρόκειται και να ταυτιστεί. Στη συνέχεια ε, εθελήσαμε να ε, εμπλέξουμε και τους πολίτες και τους χρήστες ε, όχι μόνο εκείνους που έχουν συμφέρον ή ενδιαφέρονται, αλλά ε, τους προσεγγίσαμε, αλλά και επειδή έχουν πολύ μεγάλη γνώση. Εκεί ζουν οι άνθρωποι και εργάζονται και ξέρουν πολύ καλύτερα από οποιοδήποτε δημόσιο υπάλληλο την περιοχή τους. Uh, Εδώ βλέπετε αριστερά λοιπόν ένα Google Map ε, όπου καλέσαμε τους πολίτες να μας πούν ποια είναι τα προβλήματα και ποιες είναι οι αρετές και τα πλεονεκτήματα και απάντησαν περίπου χίλιοι καθημερινοί χρήστες και κάτοικοι της περιοχής. Εκείνοι εντόπισαν τα θέματα, τα προβλήματα και μας περιέγραψαν καθημερινά πώς ζούνε στην περιφέρεια αυτή. Και βέβαια χρησιμοποίησαμε και newsletter και website, πιο κλασικά εργαλεία που τα γνωρίζετε όλοι σας. Τέλος, θα ήθελα να το συνδέσω λίγο με τις πολιτικές συνοχής. Για να είμαι ειλικρινής, η πολιτική εδαφικής ανάπτυξης και η πολιτική συνοχής ε, συνδέονται με αλλά με έναν τρόπο πάρα πολύ βαρύ. Ε, θελήσαμε να ε, χρησιμοποιήσουμε ως μοχλό την εδαφική διακυβέρνηση Βλέποντας τα διάφορα έργα και τα διάφορα project και σχέδια, χρειάζεται λίγη περισσότερη βοήθεια για να γίνει το επόμενο βήμα. Επίσης είχαμε συμφωνήσει σε επίπεδο υπηρεσιών για να ε, γίνει πραγματικότητα το σχέδιό μας. Ωστόσο, η χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, διέπεται πολύ περισσότερο συχνά από πολιτικά και λιγότερο από αντικειμενικά κριτήρια. Θα πρέπει λοιπόν κάθε φορά να γίνεται συζήτηση σε πολιτικό επίπεδο. Το θέμα της εδαφικής διακυβέρνησης είναι ζήτημα αναδιανομής κονδυλίων εντός της περιφέρειας. Αυτό είναι δύσκολο χείρημα και ακαθόδες και απαιτεί ισορροπία ε, μεταξύ των διαφόρων υποπεριφερειών, επαρχιών στην επικράτειά μας και τελικά κάθε επικράτεια, κάθε έδαφος θέλει να έχει το κομμάτι της πίτας που του αναλογεί από την πίτα χρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα τελευταία τρία χρόνια που δραστηριοποιούμε σε αυτά τα ζητήματα το συγκεκριμένο σχέδιο ε, ε, στη χρηματοδότηση υπάρχει πρόβλημα, ιδιαίτερα για την περιφερειακή διακυβέρνηση. Θα πρέπει πρώτα να καταλάβει κανείς ότι οι περιφέρειες και η περιφερειακή διοίκηση μπορούν από μόνες τους να κάνουν πολλά πράγματα. Αυτό το καταλάβαμε όταν αρχίσαμε το πρόγραμμα και κάνουμε αυτά που ξέρουμε να κάνουμε. Άρα ποια είναι η προστιθέμενη αξία που μπορεί να φέρουν τα ευρωπαϊκά κονδύλια μπορούν να υποστηρίζουν έργα που ξεπερνούν τα τετριμένα και τα συνηθισμένα. Που είναι κάπως ευρύτερα, ε, γενικότερα και σε περιφέρειες που υπάρχουν ε, διαφορετικές ε, γεωγραφικές ε, ενότητες που συμμετέχουν. Αυτή είναι η εμπειρία μας και ίσως και μια συμβολή από πλευρά μου. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ και ευχαριστώ πάνω απ' όλα για την πολύ ειλικρινή σας παρουσίαση και την εμπειρία σας που είναι πολύ πλούσια. Ποιος θέλει το λόγο τώρα αγαπητοί συνάδελφοι. Έχετε απορίες. Ο κύριος Βανίλ Στερόι. Ευχαριστώ. Και ευχαριστώ για τη διοργάνωση αυτού του σεμιναρίου. Μόλις ξεκινούμε μία, τις εργασίες για μία έκθεση της πρωτοβουλίας με το θέμα αυτό. Και χαίρομαι που ήρθατε για να μας δώσετε και συστροφή για σκέψη και στοιχεία που θα συμπεριληφθούν και σε αυτήν την έκθεση πρωτοβουλίας. Προσπαθώ να συνδυάσω αυτά που άκουσα και καταλήγω σε κάποιες αντιφάσεις. Για να δούμε την προστιθέμενη αξία των ευρωπαϊκών κινήτρων και των ευρωπαϊκών κονδυλίων. Έχουμε αφενός τους φλαμανδούς εκπροσώπους που μας λένε ότι η προστιθέμενη αξία των ευρωπαϊκών παρεμβάσεων δεν είναι εμφανής, πρέπει να την ψάξει κανείς, είναι επαξής η διαδικασία αν όμως επαχθείς μια διαδικασία, γιατί να την προωθήσουμε. Απ' τη μια λοιπόν βλέπουμε αυτή την εμπειρία α, της α, εδαφικής διακυβέρνησης που είναι μακροχρόνια και ο πρώτος ερευνητής μας είπε ότι για τη θεματική συγκέντρωση είχαν κάποιες επικρίσεις, μα η θεματική συγκέντρωση ακριβώς είναι η λύση σε αυτή την επαχθή κατάσταση. Αυτή είναι η λύση στο πρόβλημα της επαχθούς διαδικασίας. Το γεγονό ότι δίνουμε κονδύλια στι περιφέρειες να κάνουν ό,τι θέλουν και να δώσουν αυτή την ε, εδαφική, ε, εδαφική προσέγγιση, αλλά να ε, επικεντρωθούμε σε αποτελέσματα για ολόκληρη την Ευρώπη. Γιατί αυτό μας ενδιαφέρει είναι η ανάπτυξη και η απασχόληση. Όχι να βελτιώσουμε την διακυβέρνηση των πόλεων. Κάθε πόλη έχει τη δική της διακυβέρνηση. Είχαμε κάποιες διαφορές μεταξύ της πρώτης ομιλίας και των άλλων σχολείων που ακούσαμε. Φυσικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα κάνει κάποιες επιλογές και θα εφαρμόσει αυτές τις πολιτικές. Είπατε κάτι που έχουμε συζητήσει και εμείς, ότι η έκτη έξεση συνοχής δεν έχει καλή αναλυτική παρουσίαση. Η πέμπτη έκθεση της συνοχής ήταν πολύ καλύτερη. Ενώ η έκτη δεν είναι τόσο καλή σε διαφορά την εδαφική συνεργασία. Χωλαίνει κάπω. Πού οφείλονται οι αδυναμίε τη και ποιε είναι οι διαφορέ τη πέμπτη και τη έκτη έκθεση συνοχή. Η πρόεδρο ε, ε, σε μια συνάντηση που είχε με την Επιτροπή των Περιφερειών ε, κατάλαβε ότι η Επιτροπή των Περιφερειών υιοθετεί αυτή την εδαφική προσέγγιση και μάλιστα θα συντάξει και έκθεση η Επιτροπή των Περιφερειών με αυτό το θέμα και εκεί φαίνεται ότι αυτό που βλέπετε εσείς ε, ως ε, ε, εθνικοποίηση δεν είναι κάτι καινούριο. Ίσως πρόκειται για μια επανεθνικοποίηση. Έχουμε και το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο που είναι εθνικό θέμα ή η στρατηγική για το 2020. Λέτε ότι έχει ιδιαίτερα εθνική εστίαση. Ο κύριος Ρώσο όμως στην έκθεσή του εξακολουθεί να πιστεύει στην περιφερειακή διάσταση της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για το 2020. Ποιο είναι κατά τη γνώμη σας το μέλλον της εδαφικής συνοχής. Είναι δύσκολη και παχθής η διαδικασία και αν θεωρείτε ότι είναι υπερβολικά μπερδεμένοι, θα πρέπει να επανέλθουμε και να ενισχύσουμε την εδαφική συγκέντρωση, την τομεακή οικονομική συγκέντρωση. Επίσης, για τα αριθμητικά στοιχεία. Έχουμε ε, από τον ΩΣΑ μια ολόκληρη βιβλιογραφία με διαφορετικές ε, καταστάσεις. Είπατε όμω σε μερικές χώρες 10% ε, των χρημάτων ξοδεύονται από τις περιφέρειες στις περιφέρειες στην Ελλάδα μπορείτε να μας πείτε ή θεωρείτε ότι μία μεγαλύτερη ανάμειξη, μεγαλύτερο τμήμα του προπολογισμού και πιο ολοκληρωμένη περιφερειακή πολιτική αποφέρει περισσότερους καρπούς και δημιουργεί περισσότερες θέσεις απασχόλησης. Γιατί. Καλά δεν μιλάμε για την ε, διακυβέρνηση, αλλά δεν έχουμε περισσότερη ανάπτυξη και απασχόληση στο μέλλον θα μείνουμε σε μια αποτελεσματωμένη κατάσταση. Ποια είναι η, η λύση. Πιο αποκεντρωμένη διαχείριση όπως στη Γερμανία και ποιο είναι το αποτέλεσμα. Ερωτήσεις περισσότερο θέτω παρά έχω απαντήσει. Ευχαριστώ. Ξέρω ότι είστε έτοιμοι να απαντήσετε σε απορίε του κύριου Βανίστε αλλά συγκεντρώσουμε πρώτα όλε τι ερωτήσει και μετά θα ακούσουμε του εμπειρογνώμονέ μα για τι απαντήσει. Ο κύριο Έτεριτ έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Εγώ έχω πιο συγκεκριμένες ερωτήσεις. Ακούσαμε ομιλίες για την εδαφική διακυβέρνηση και για το σχετισμό της με την πολιτική συνοχής. Εμένα με ενδιαφέρουν τα West Midlands στην Αγγλία, από αυτή την εκλογική περιφέρεια εκπροσωπώ. Τώρα σκοπεύουμε να έχουμε μια συνδυασμένη αρχή για ολόκληρο τα West Midlands. Συνεχίζεται βέβαια η συζήτηση για το θέμα αυτό και είναι αρκετά επίμαχη και φλέγουσα η συζήτηση. Χρειάζονται ε, μια τέτοια συνδυασμένη αρχή θα καλύπτει 7 δημοτικά συμβούλια και 3 πόλεις για το σύνολο των West Midlands. Κατά τη γνώμη σας, ποιο θα ήταν ένα θετικό βήμα προς μια συνοχή, πολιτική συνοχή και εδαφική διακυβέρνηση. Επιπλέον, θα ήταν δυνατό ένα ή δύο από τα δημοτικά συμβούλια της ευρύτερης περιφέρειας να συζητήσουν θέματα που συζητούμε και εμείς στη δική μου περιοχή τώρα. Για να ακούσουμε και από τους ειδικού ποια είναι η γνώμη τους για το θέμα της συνοχής. Γιατί, όπως είπαμε, σε μια συνδυασμένη αρχή ίσως δεν υπάρχει μια λύση για όλους. Ίσως εκεί θα πρέπει να εφαρμόσουμε περισσότερη ευελιξία και περιθώριο ελιγμών. Θεωρείται λοιπόν ότι μια συνδυασμένη αρχή σαν αυτή των West Midlands, όπω συζητάτε τουλάχιστον τώρα, θα βοηθήσει στο θέμα τη ευρωπαϊκή εδαφική διακυβέρνηση. Ευχαριστώ κύριε Στέλλερ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Καταρχά θέλω να ευχαριστήσω και του εμπειρογνώμονε μα για τα όσα μα είπαν και μα παρουσίασαν. Μα έδειξαν μια πολύ χρωμή εικόνα και την ποικιλία που επικρατεί στην Ευρώπη σε ό,τι αφορά τη διοίκηση και την αυτοδιοίκηση και πώς έχει ο πολιτικός διαχωρισμός στα διάφορα κράτη-μέλη. Είναι πραγματικά πολύχρωμη εικόνα, υπάρχουν πολλές διαφορές από χώρα σε χώρα. Έχω ασχοληθεί στο παρελθόν με την αυτοδιοίκηση και γνωρίζω ότι οι πολίτες εκεί κινητοποιούνται και δραστηριοποιούνται και πολιτικά. Αυτό είναι το επίπεδο που τους ενδιαφέρει. Όταν είναι καθημερινά τα προβλήματα και στη βόρτα του σπιτιού τους. Από εκεί ξεκινάει η πολιτική. Και όσο προχωρούμε και ανεβαίνουμε σε επίπεδο διακυβέρνησης, τόσο περιπλέκονται τα πράγματα και τόσο πιο δύσκολα είναι να εξηγηθούν στον καθένα και να τον κινητοποιήσουν. Το υψηλότερο πολιτικό επίπεδο που έχουμε είναι το ευρωπαϊκό, που είναι ακόμα πιο περίπλοκα και πιο θολά τα πράγματα και σκοτεινά. Οπότε και γι' αυτό το λόγο η περιφερειακή πολιτική και η πολιτική συνοχή εφευρέθη κάποτε για να δημιουργήσει αυτή τη γέφυρα και να κλείσει ο κύκλος και να συναντήσει ξανά η ευρωπαϊκή πολιτική των πολίτη. Και με την ευρωπαϊκή υποστήριξη και τα ευρωπαϊκά κονδύλια να φανεί η Ευρώπη στις περιφέρειες και τις υποπεριφέρειες ε, με έργα που θα μιλάνε στους πολίτες και που δεν θα ήταν δυνατόν να κατασκευαστούν με ιδίους πόρους ή που δεν είναι δυνατόν. Εγώ μιλώ για το Ανατολικό Βερολίνο και τα ανατολικά κρατήδια της Γερμανίας και αν δω τη διαφορά ε, που έχουν με τη Δυτική Γερμανία, με το Δυτικό Βερολίνο, χρειάστηκαν 15 χρόνια και πλέον ε, για να ε, έρθουν κοντά οι περιφέρειες. Απέδωσε όμως αυτή η προσπάθεια, αλλά χρειάστηκαν 15 χρόνια. Λοιπόν, τώρα έχουμε τη νέα προγραμματική περίοδο και διαπιστώνουμε το εξής. Τις τελευταίες 15 μέρες είχα την ευκαιρία να συζητήσω με ανθρώπους που είναι πάρα πολύ ενεργοί στην περιφερειακή πολιτική και την πολιτική συνοχής και εργάζονται για τα διάφορα μόσπονδα κρατήδια της Γερμανίας και είναι ο σύνδεσμος ανάμεσα στο ευρωπαϊκό επίπεδο, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τους επιτόπου ε, φορείς στις πόλεις και στα ομόσπονδα κρατήδια. Και τι ακούω από αυτούς, ότι στο μεταξύ η πολιτική συνοχής σχεδόν ε, δεν μπορεί να υλοποιηθεί στην πράξη για τους ενδιαφερομένους. Μιλάμε συνεχώς για απλούστευση, για άρση γραφειοκρατίας και τώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεσπίζει κανόνες για τις περιφέρειες και για τις ενδιάμεσες δομές που είναι τόσο ε, αδιαφανείς ε, και χρειάζεται τόσο πολύ ευθύνη που σηκώνουν τα χέρια ψηλά οι άνθρωποι επιτόπου και σου λένε εγώ δεν μπορώ να τα επιμιστώ όλα αυτά. Και ρωτώ, αυτό είναι εσκεμμένο. Για ποιο λόγο έχουν περιπλακεί τόσο πολύ οι καταστάσεις και οι διαδικασίες. Διότι αν εμείς δεν μπορούμε τη διορθωτική πολιτική και την πολιτική συνοχής να την ασκούμε ως περιφερειακή πολιτική, εάν κράτη χρησιμοποιούν κονδύλια από τα ταμεία συνοχής για τις κρατικές του δημόσιες επενδύσεις, τότε για μένα η πολιτική συνοχής και η διαρθρωτική πολιτική στερείται την ψυχή της, γιατί της την κλέβουν και ε, δεν ξέρω αν θα πρέπει να συνεχιστεί καν. Και σε ό,τι αφορά τη θεματική συγκέντρωση, αγαπητέ Λάμπερτ, Βανίστε ροή διαφωνώ κάθετα. Βεβαίως χρειαζόμαστε θεματική συγκέντρωση και θα πρέπει να χρησιμοποιούμε με νόημα τα κονδύλια και να μην τα σπαταλάμε, να μην τρέχουμε ας πούμε καλοκαιριάτικα μέσα στην τάδα να ποτίζουμε λιβάδια. αλλά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δίνει στις περιφέρειες κάποιες οδηγίες κάποιες υποδείξεις για τις θεματικές συγκεντρώσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δηλαδή τα απαγορεύει και όχι αυτό που θεωρούν χρήσιμο και σκόπιμο οι ίδιες οι περιφέρειες. Όταν συζητούσαμε τους κανονισμούς, πριν λάβουμε τις αποφάσεις, είχαμε αυτή την παράκληση από τις περιφέρειες, την οποία διαβιβάσαμε και διευρύναμε τον κατάλογο των θεμάτων. Από ό,τι φαίνεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη συζήτηση με τις περιφέρειες και εκείνους που διαχειρίζονται τα κονδύλια το έχουν ξεχάσει. Θεωρεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι μπορεί να επαγορεύει σε μια περιφέρεια τι είναι σημαντικό και χρήσιμο και απαραίτητο για τους στόχους τους δικούς της, της Κομισιόν. Επίσης, ό,τι αφορά την αστική ανάπτυξη τους Δήμους, ε, εκεί που συνενώνονται ε, κάποιες ε, αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης για να κάνουν κοινά προγράμματα με ευρωπαϊκή υποστήριξη, κατακλείζονται με νέες απαιτήσει, γραφειοκρατία, ε, σχολαστικές ε, οδηγίες, υποδείξεις. Υπό την επικεφαλίδα καταπολέμηση της διαφθοράς βέβαια, αλλά πολύ συχνά είναι τόσο μικρά τα έργα που δεν τίθεται θέμα διαφθοράς. Νομίζω θέλει πολύ μεγάλη προσοχή εδώ να μην ε, φορτώσουμε πάρα πολύ με κανόνες ένα καλό πεδίο πολιτικής που αντανακλά αυτή την ποικιλομορφία και την πολυχρωμία στην Ευρώπη γιατί διαφέρουν οι περιφέρειες. Θέλει προσοχή αυτό. Μέχρι τώρα είχαμε κονδύλια για τη διαρθωτική και την πολιτική συνοχή και θέλαμε να ενδυναμώσουμε τις περιφέρειες, να χειραφετηθούν, να έχουν την ευκαιρία με ευρωπαϊκή υποστήριξη να διαχειρίζονται τα ζητήματά τους και τα ενδιαφέροντά τους με τη λύση που εκείνες θεωρούν ε, σκόπιμη. Τώρα θέλει προσοχή, μην τυχόν και με τέτοιες μεθόδους που σας περιέγραψα ε, καταστρέφονται. Γιατί όταν συνθηκολογούν οι περιφέρειες, καταθέτουν τα όπλα και σηκώνουν τα χέρια ψηλά και δεν συμμετέχουν στα διαστρωτικά προγράμματα ή στις υποδομές, τότε μετά το 2020 δεν χρειάζεται πια να το συζητούμε καν. Ελπίζω να μην είναι πρόθεση αυτό εκείνων που ασκούν τη διοίκηση. Και ε, ασχολούνται με την περιφερειακή και την υποπεριφερειακή στήριξη. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και εγώ πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά και πάρα πολύ περιστατωμένα. Είναι το πρώτο τέτοιο εργαστήριο που κάνουμε στην Επιτροπή μας. Καλό είναι όμως να ασχολούμαστε σε βάθος με ένα θέμα, μεγάλη καινοτομία και η δική μου πολιτική ομάδα ήταν εκείνη που ζήτησε τη μελέτη ε, για την εδαφική διακυβέρνηση και έχουμε μάθει πολλά ήδη για τις εμπειρίες σας και για τις ιδέες σας. Έχω δύο σύντομες ερωτήσεις. Ερώτηση πρώτη προς τον κύριο Μπέμε και την κυρία Τσίλμερ κυρίως. Πολύ συχνά τονίσατε ότι δεν υπάρχει μία ενιαία προσέγγιση για όλους, ένα μέγεθος ας πούμε που να κάνει σε όλους, αλλά έχετε εντοπίσει κάποιους παράγοντες που οδηγούν στην επιτυχία ή κάποιες βέλτιστες πρακτικές. Να μας δώσετε ένα παράδειγμα για καλή διακυβέρνηση και ένα άλλο για κακή διακυβέρνηση. Ποια είναι τα κριτήρια που χρησιμοποιείτε και ποιες οι εμπειρίες σας. Και δεύτερη ερώτησή μου αφορά τη χειραφέτηση των τοπικών φορέων, ενδυνάμωση, αυτό το empowerment, το είπαν και οι προλαλήσαντες. Και ο κύριος Ρενέ Φαντερλέκ από τη Φλάνδρα, με αυτή την υφάλια ανάλυση ότι τα κονδύλια των διαρθρωτικών ταμείων χορηγούνται με βάση πολιτικά κριτήρια και λιγότερο αντικειμενικά, με βάση το έργο. Γι' αυτό το λέμε εμείς από μια επιτροπή που μιλάει για θεματικούς στόχους, για την προστασία του κλίματος, για την αστική ανάπτυξη κτλ. Να έχουμε στοχευμένες παρεμβάσεις και προσπαθούμε να τις υλοποιούμε. Έχετε συστάσεις να μας κάνετε υποδείξεις, προτάσεις για το τοπικό επίπεδο και το περιφερειακό, πώς μπορούμε να βοηθήσουμε για αυτό το empowerment. Το ξέρω ότι είναι πάρα πολύ ασαφής η ερώτησή μου ε, και τώρα Έχασα και τον ήρμο, πώς το λένε αυτό στα γερμανικά, για το empowerment. υπάρχει τεχνογνωσία για τη σωστή ε, υλοποίηση όλων αυτών των προγραμμάτων. Ο κόσμος τόπου ξέρει τι χρειάζεται και τι μπορεί να αποκομίσει από τα διευθυντικά ταμεία. Ευχαριστώ. Μόγκοβιτς. Hvala lepa za to poročilo in za današnjo eh, σας ευχαριστώ πολύ. Πολύ χρήσιμη αυτή η συζήτηση και για την έκθεσή μας. Πολύ σημαντική. Έχω μακροχρόνια εμπειρία, 13 χρόνια, ως δήμαρχος ε, πριν γίνα, πριν εθνικός βουλευτής και κατόπιν ευρωβουλευτής. Έχω εργαστεί λοιπόν πακρόν στις ε, περιφερειακές ε, και τοπικές ε, κοινότητες, στην τοπική αυτοδιοίκηση και από την εμπειρία μου αυτή έχω αποκομίσει την ακράδαντη πεποίθηση ότι η καλή οργάνωση σε τοπικό επίπεδο είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την σωστή διακυβέρνηση και σε εθνικό επίπεδο. Και Βλέποντας την τέταρτη και πέμπτη διαφάνεια, διαπιστώνω ότι είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι οι διαστάσεις των τοπικών φορέων και περιφερειακών φορέων είναι σημαντικές τα μεγέθη, αλλά δεν έχουν άμεση σχέση με την ανάπτυξη, με το επίπεδο της ανάπτυξής τους. Στην ε, πέμπτη διαφάνεια το σημαντικό στοιχείο είναι η επικουρικότητα. Φαίνεται ότι οι χώρες με ανεπτυγμένο τοπικό επίπεδο είναι αυτές που έχουν μεγαλύτερη ανάπτυξη και σε εθνικό επίπεδο. Θα πρέπει λοιπόν ε, να τονίσουμε και τις λειτουργικές σχέσεις που ισχύουν και πώς συνδέουμε τις ε, τοπικές κοινότητες και τις περιφέρειες μεταξύ τους. Έτσι θα αποκτήσει ενδιαφέρον η συζήτηση. Και πολύ γρήγορα θα βρούμε και κοινά σημεία. Όταν έχουμε δηλαδή απευθείας συνεννόηση με τους άμεσα ενδιαφερομένους. Πέρα λοιπόν της οργάνωσης σε εθνικό επίπεδο θα πρέπει να δούμε και την οργάνωση και τον τρόπο εφαρμογής των σχεδίων. Γιατί στην πολιτική συνοχής πολύ συχνά σε μια περιοχή, σε μια περιφέρεια από στατιστική άποψη είναι δύσκολο να εφαρμόσουμε κάποια σχέδια. Γι' αυτό θα πρέπει να επικεντρωθούμε στο σημείο αυτό και να ασχοληθούμε περισσότερο με το περιεχόμενο για να εφαρμόσουμε στο μέλλον μια πολύ καλύτερη πολιτική συνοχής. Γιατί μια τέτοια πολιτική θα βοηθήσει την καλύτερη συνεργασία και επαφή των ανθρώπων αλλά και των περιφερειών για συγκεκριμένα σχέδια που θα έχουν και χειροπιαστά αποτελέσματα. Και έτσι θα φανεί και η προστιθέμενη αξία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα είμαι σύντομος γιατί ε, τελειώνει και ο χρόνος. Μια σύντομη ερώτηση για την ε, εδαφική διακυβέρνηση που κατά τη γνώμη μου δεν είναι αυτός ο σκοπός. Ε, ήταν ε, εξάλλου νομίζω το θέμα ε, που έθιξε και ο Λάμπερτ Φανίστερ Ρόι. Πώς μπορείτε να συμβάλλετε πραγματικά σε μια στρατηγική Ευρώπη 2020 που εστιάζει στην απασχόληση και τη βιώσιμη μάλιστα απασχόληση. Και δεύτερη ερώτηση, γιατί έχω αυτή εδώ την έκθεση. Ό,τι σχετίζεται με τις στρατηγικές της ευθυούς ειδίκευσης. Τι μπορείτε να μας εξηγήσετε όσον αφορά τα, τις σωστές δεξιότητες ε, για την ε, ε, περιφερειακή διακυβέρνηση και πώς δηλαδή θα μπορέσουν πραγματικά να φτιάξουν μια στρατηγική καινοτομία που θα βασίζεται στην ευφυή ειδίκευση. Σας ευχαριστώ πολύ για την ερώτησή σας. Αυτό είναι το τμήμα της ερώτησης που ήθελα και εγώ να θέσω γιατί συνεχίζεται η συζήτηση αυτή ανάμεσα στους δύο μας, διότι εγώ είμαι υπέρμαχος της εδαφικής διάστασης της πολιτικής συνοχής, διότι πιστεύω πράγματι ότι η εδαφική προσέγγιση είναι αυτή που μας δίνει τα αποτελέσματα πιο κοντά στους πολίτες της Ευρώπης. Από την άλλη πλευρά, Έχουμε μια άλλη εικόνα της εθνικοποίησης, όπως αναφέρατε, σε περισσότερα προγράμματα. Σας ευχαριστώ λοιπόν για τις παρουσιάσεις. Υπάρχουν άλλες ερωτήσεις? Όχι. Οπότε μπορείτε να απαντήσετε παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ για τις πολύ ενδιαφέρουσες και πλούσιες ερωτήσεις. Εγώ θα ξεκινήσω και μετά ελπίζω πως η Σαμπίνε θα συμπληρώσει διάφορα. Να ξεκινήσω με αυτό που είπε ο κύριος Φανίστελ Ρόι, ότι πρέπει να είμαστε σαφείς. Από τη μια πλευρά όταν μιλάμε για ε, επίπεδο project, έχουμε ένα παράδειγμα από τη Φλάνδρα που λέει ότι έχουμε ένα project και τη διαχείρισή του και αυτό είναι εξαιρετικά δύσκολο εγχείρημα. Ε, πρέπει να δούμε πως ε, οι κανονισμοί είναι πολύ πιο αυστηροί ε, και χρειάζεται συγκεκριμένη δεξιότητα για να μπορεί να το κάνει αυτό κάποιος. Ε, εμείς δεν είδαμε πραγματικά τα προγράμματα λέξη προς λέξη. Εμείς είδαμε κάπως γενικότερα και από πιο ψηλά ε, το πώς θα μπορούσε να λειτουργήσει. Τώρα, αν εξετάσουμε πώς άλλαξε τα πλαίσια πολιτικής, θέλαμε να δούμε αν αυτές οι αλλαγές οδηγούν σε περισσότερη δημοκρατική διακυβέρνηση ή όχι. Και έπειτα σε αυτό το τμήμα Θέλαμε να κάνουμε και μια εσωτερική συζήτηση όσον αφορά τη θεματική προσανατολισμό και το προσανατολισμό στα αποτελέσματα. Αυτό μας αρέσει γιατί σημαίνει ότι εστιάζουμε σε αυτό το θέμα, αλλά μειώνεται ο αριθμός των φορέων που συμμετέχουν. Υπάρχει μια αντίφαση δηλαδή στους στόχους. Ανάλογα με το τι αναζητείς θα πρέπει να ενεργήσεις προς τη μια κατεύθυνση ή προς την άλλη. Για την αδερφική διακυβέρνηση θα έπρεπε να εφαρμόσουμε αυτήν την ε, ε, στρατηγική, αλλά είχαμε και εσωτερικέ συζητήσεις και δυσκολίες. Ανάλογα λοιπόν με τις προτεραιότητες θα δώσεις περισσότερο βάρος στο ένα ή στο άλλο στοιχείο για την Ευρώπη 2020. Δεν περιλαμβάνει πολύ έντονη διάσταση δαφικής διακυβέρνησης ε, στην ε, στην επεξεργασία, αλλά στην εφαρμογή του, το πρόγραμμα αυτό εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τα όσα γίνονται επί τόπου. Είναι μια δυναμία του εγγράφου, ε, ώστε να μπορέσουν δηλαδή να οικειοποιηθούν οι άνθρωποι σε τοπικό επίπεδο τα προγράμματα. Η Ευρώπη 2020 υποτίθεται ότι είναι το κοινό μας όραμα των Ευρωπαίων και αυτά τα έγγραφα πρέπει να καλύπτουν και αυτές τις διστάσεις. Τώρα εγώ δεν έχω κάποιο σχέδιο για το πώς θα λυθεί αυτό το θέμα. Αλλά υπάρχει τρόπος να συμμετέχουν τοπικοί και περιφερειακοί ε, φορείς στην αναθεώρηση αυτών των εγγράφων ώστε να έχουμε μια ένα ισχυρότερο κοινό όραμα και μια ισχυρότερη δαφική διακυβέρνηση. Πράγμα το οποίο μετά θα μεταφραστεί και στην εφαρμογή του εν λόγω εγγράφου αργότερα. Προσπαθήσαμε λοιπόν να δούμε από αυτή την προοπτική της εδαφικής διακυβέρνησης αυτό το θέμα και μετά υπάρχουν διάφορα σημεία που μπορούμε να συζητήσουμε από διαφορετική οπτική γωνία και μετά βεβαίως θα φτάσουμε σε διαφορετικό συμπέρασμα. Α, α, α, τώρα βέβαια το επίπεδο λήψης αποφάσεων είναι αυτό που θα αποφασίσει τι θα γίνει τελικά. Υπήρξε και το ερώτημα των Δυτικών Midland και ο συνδυασμός των αρχών σε ένα είδος πιο περιφερειακής αρχής και αν αυτό στηρίζει την εδαφική διακυβέρνηση ή όχι. Πρέπει να σας πω ότι δεν ξέρω τι ακριβώς γίνεται στα Δυτικά Midlands, οπότε ε, εγώ θα ξεκινούσα από το εξή. Αυτό που είπε ο συνάδελφος από τον ΟΣΑ. Οι λειτουργικές μονάδες σε ποιο βαθμό μπορεί να καλύψει όλους τους τους Δήμους τους οποίους αναφέρετε εσείς και πώς μπορούν αυτοί να συνδυαστούν και ως λειτουργική μονάδα πώς θα μπορέσει να συνεργαστεί ώστε να προσεγγίσει τις αναπτυξιακές ανάγκες της περιοχής ώστε να μπορέσουν δηλαδή να συνδυαστούν. Θα πρέπει δηλαδή να φροντίσουμε ώστε να βρούμε τις καλύτερες προϋποθέσεις για να προσεγγίσουμε ε, την ε, δευτική κυβέρνηση. Τώρα αν θα τυποποιηθεί όχι το θέμα, ε, αυτό συζητάται στην Ευρώπη. Προσπαθούμε να δουλέψουμε σε διάφορα επίπεδα. Υπάρχουν διαφορετικοί τρόποι για να προσεγγίσουμε το θέμα. Ένα άλλο σημείο για την καλύτερη πρακτική και τα κριτήρια επιτυχίας. Υπάρχουν πολλές ενδιαφέρουσες καλές πρακτικές. Οι βέλτιστες πρακτικές λίγο διστάζουν να το πω, αλλά πάντως αν μιλάμε γενικά για την εδαφική δικυβέρνηση, θα έλεγα ότι βασίζεται στις ε, αναπτυξιακές ανάγκες όπως είπα. Αυτή είναι η προϋπόθεση για να είναι καλή η διακυβέρνηση και αυτό σημαίνει τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων και εμπληκωμένων φορέων, να υπάρχει ένα κοινό όραμα, κάτι το οποίο έχετε επεξεργαστεί από κοινού. Και νομίζω δύο, παράδειγμα που, δύο παραδείγματα που μου ήρθαν στο μυαλό. Το ένα αφορά την περιφέρεια της Στοκχόλμης, όπου υπάρχουν πολλά θέματα αναπτυξιακά λόγω της μεγάλης εξουσίας του τοπικού επίπεδου. Άρα λοιπόν αντιμετωπίζονται στο τοπικό επίπεδο, αλλά για να λυθούν πρέπει να προσεγγιστούν σε περιφερειακό επίπεδο, γιατί αυτό που συμβαίνει στον ένα Δήμο επηρεάζει και τον άλλον. Το περιφερειακό επίπεδο δεν είναι πολύ δυνατό όσον αφορά τις αρμοδιότητές του. Και κάποιος στην περιφέρεια της Στοκχόλμης είπε μπορούμε να καλέσουμε τους υπόλοιπους σε διάλογο και έτσι να γίνει κάτι πιο ενίδη ε, εν παιχνιδιού. Το αποκάλεσαν και παιχνίδι ώστε επειδή έχουν 7 διαφορετικά επίπεδα διακυβέρνησης να μπορέσουν να συντονιστούν και να εντοπίσουν λύσεις και προκλήσεις σε όλη την περιφέρεια. Κάλεσαν λοιπόν όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς να συγκεντρωθούν, να παίξουν στο ίδιο παιχνίδι, να δουν στην πράξη πώς λειτουργούν τα πράγματα και πώς επηρεάζουν οι πράξεις των ενός των άλλων και τούμπαλιν. Και στις αρχές ο κόσμος δεν τα έπαιρνε όλα αυτά σοβαρά, αλλά σιγά σιγά έρχονται να συνειδητοποιούν ότι έρχονται να μαθαίνουν και πράγματα για το πώς ε, είναι αλληλένδετα όλα ανάμεσα στα διάφορα επίπεδα διακυβέρνησης και τις διάφορες πολιτικές. Αρχίσαν λοιπόν να αλλάζουν και έτσι προσέθεσαν άλλη μια γραμμή προτεραιότητας στο IOP. Υπήρξαν δηλαδή συνέπειες και αλλαγές. Περισσότερο όμως πρόκειται για τεχνικές, για το πώς μπορεί κανείς να δημιουργήσει μια πλατφόρμα για να αποφύγει τα παιχνίδια εξουσίας ή αρμοδιοτήτων. Κάτι ακόμα είναι πολύ ενδιαφέρον από τη Τιμισοάρα της Ρουμανίας. Και η Ρουμανία δεν είναι γνωστή για την ισχυρή διακυβέρνηση. Δεν είχαμε προβλήματα με τους μετανάστες που έφταναν στη Τιμισοάρα, κυρίως από χώρες που δεν είναι μέλη της Ένωσης και αντιμετώπιζαν πολλά πολλά προβλήματα ε, στην δημόσια διοίκηση γιατί δεν μπορούσαν να την προσεγγίσουν. Έτσι την όριζαν. Υπήρξε μια μήκη όμω που χρόνια και χρόνια προσπάθησε ξανά και ξανά να συγκεντρώσει όλους τους αρμόδιους φορείς ώστε να βρεθεί μια λύση για το πώς θα μπορούσαν να διευκολυνθούν οι ζωές αυτών των μεταναστών και πώς θα μπορούσαν να έχουν πρόσβαση στην παιδεία, στην απασχόληση και ούτω καθεξής. Τελικά τα κατάφεραν τόσο καλά όλοι αυτοί από την ΜΚΟ. Δημιουργήθηκαν και διάφορες ενδιάμεσες δομές και αντιγράφηκε σε άλλα μέρη της Ρουμανίας και μάλιστα φτάσαν να συζητούν το εναλλαγή του εθνικού νομικού συστήματος ώστε όλα αυτά να λειτουργούν πιο ομαλά. Μικρές λεπτομέρειες δηλαδή που όμως στην πράξη ε, ε, έπρεπε να, στην πράξη έπρεπε να απλοποιηθούν κάποιες πολύ χρονοβόρες και βαριές διαδικασίες. Πρέπει δηλαδή να μπορέσεις να λειτουργήσεις με βάση τα όσα υπάρχουν. Και αυτό είναι ένα μόνιμο πρόβλημα. Πώς δηλαδή θα μπορέσουν οι άνθρωποι που έχουν την ιδέα και που βρίσκονται επί τόπου να τα καταφέρουν. Πώ θα τους δώσουμε τη δυνατότητα να τους βοηθήσουμε. Τουλάχιστον εγώ δεν έχω δει καμία πραγματική παρότρινση. Περισσότεροι ξεκινούν μειώνοντας τον αριθμό των εμποδίων. Όπως είπαν οι, οι κυρίες της ΜΚΟ από τη Ρουμανία, είπαν ότι αν δεν μπορείς την πόρτα, πρέπει να, να μπεις από την πόρτα σε ένα κτίριο, πρέπει να μπεις από το παράθυρο. Ε, πρέπει δηλαδή κάτι να αλλάξει και να ξαναπροσπαθήσει. Το ίδιο και έγινε και στη Στοκχόλμη. Αυτό που ξεκίνησε αυτό το παιχνίδι έπρεπε να καταπολεμήσει τη γελιοποίηση που δέχτηκε στην αρχή. Ε, γιατί το πήγε σαν να ήταν παιχνίδι και αστιάκι. Και σιγά σιγά να αλλάξουν. Δηλαδή πρέπει να μπορέσουν να ενθορυνθούν, να παροτρινθούν. Ε, πάντως ένα θεσμικό όργανο δύσκολα θα μπορούσε να κάνει τέτοια πράγματα. Η καλή οργάνωση τοπικό και περιφερειακό επίπεδο φυσικά εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το εθνικό πλαίσιο. Εννοείται. Αλλά οι κυβερνητικέ διαδικασίε δεν περιορίζονται μόνο στο δημόσιο τομέα, αλλά και σε μη δημόσιου φορεί. Και έχουμε ευρύτερη εδώ σκοπιά. Και τώρα, σε ό,τι αφορά την ευφυή ειδίκευση, δεν το εξετάσαμε στη συγκεκριμένη έκθεση, αλλά το θέμα αυτό συζητάται ευρέω. Και αυτή τη στιγμή έχουμε πολλές στρατηγικές ευθείους ειδίκευσης που είναι λίγο copy-paste, απλή αντιγραφή μεταξύ των διαφόρων περιφερειών. Πάντως οι καλές σχετίζονται με τις τοπικές ιδιαιτερότητες. Θα πρέπει να δούμε τις προϋποθέσεις για την καινοτομία και τους τομείς που δίνουν μια στιβαρή βάση για κάτι τέτοιο. Και φυσικά χρειαζόμαστε και ενδιαφερομένους ε, για να αναλάβουν αυτό το θέμα. Είναι στη μόδα αυτά τα θέματα της ευθείου ειδίκευσης. Είχαμε μια Ιταλική περίπτωση, αν δεν κάνω λάθος, ένα Ιταλικό παράδειγμα, όπου κάποιοι επένδυσαν ε, στη γεωργία. Αυτό βέβαια δεν είναι ευφυής ειδίκευση, αλλά ε, ειδικεύτηκα τόσο πολύ σε ένα συγκεκριμένο τομέα της γεωργίας, που τώρα είναι ε, Παγκοσμίω ε, γνωστή σε ό,τι αφορά την προμήθεια συγκεκριμένων κλάδων. Το θέμα είναι να βρει, βρει κανεί μία δίωδο προ την ευθύ δίκευση. Αυτά και ελπίζω να με συμπληρώσει η συνάδελφο ε, η Σαμπίνε. Θα προσπαθήσω, αν και ήταν αρκετά πλήρη η απάντηση και κάλυψε πολλέ ερωτήσει. Εγώ θα συμπληρώσω κάποια μικρά κενά που έμειναν. Σε ό,τι αφορά τη θεματική συγκέντρωση, ναι φυσικά το συζητήσαμε και είπαμε δεν είναι κακή και όπως είπε ο κύριος Τσέλερ, αν συγκεντρώνουμε κονδύλια σε συγκεκριμένες τοπικές ανάγκες, είναι πολύ καλύτερο από το να λέμε πρέπει να πληρείτε την ΑΒ προϋπόθεση. Έχουμε διαφορετική προσέγγιση στη θεματική συγκέντρωση που χρειάζεται. Ρωτήσατε ποια είναι η σχέση μεταξύ της παραγωγής και του φεδεραλισμού. Όταν ακολουθούμε την αρχή της επικουρικότητας, που έχει λόγο που υπάρχει, δεν είναι για πλάκα, θέλει να φέρει η επικουρικότητα την πολιτική κοντά στον κόσμο και να πραγματοποιεί να αναλαμβάνει δράσεις εκεί που χρειάζονται και που είναι κατάλληλες. Δεν είναι ότι πάντα είναι απαραίτητο ο φεδεραλισμός ή η καλύτερη προσέγγιση, ο φεδεραλισμός ή η τοπική η η τοπικη προσέγγιση η επικουρικότητα θα πρέπει να μπορεί να παρέχει τις δράσεις στο επίπεδο που χρειάζεται, όχι πάντα στο τοπικό. Γιατί αν δεν υπάρχει θεσμική ικανότητα, αν δεν υπάρχουν κονδύλια, αν δεν υπάρχει κατάλληλη οργάνωση και αν δεν πληρούν περισσό... πολλές προϋποθέσεις, τότε δεν αρκεί μόνο το τοπικό επίπεδο. Ποιοι είναι οι πιο πετυχημένοι τομείς Αναφέραμε κάτι και στην παρουσίαση για την ε, ηγετική θέση και τις διαφορές, ε, διαφορετικές πτυχές ε, θεσμικές και διοικητικές και την οργανωτική ικανότητα που είναι απαραίτητη. Νομίζω ότι στη μελέτη μας για τα σχέδια πολυεπίπεδα διακυβέρνηση για την Ευρώπη 2020 είχαμε βρει πολύ περισσότερα στοιχεία. Και μάλιστα είχαμε κάνει και ένα κατάλογο που δεν το θυμάμαι απ' έξω, αλλά υπάρχει στη σχετική μελέτη. Ρωτήστε τι γίνεται με τη χειραφέτηση των τοπικών αρχών, την ανάληψη εξουσιών σε αυτό το επίπεδο. Κάθε επίπεδο έχει το, δικό του ρόλο και, και τα υψηλά επίπεδα μπορούν να στηρίξουν τη χειραφέτηση σε χαμηλότερα επίπεδα. Βέβαια η διαδικασία αυτή είναι χρονοβόρα. Και πρέπει να αξιοποιηθούν οι ικανότητες ε, και να δείξει κανείς υπομονή και επιμονή και δεν μπορούμε να επιβάλλουμε κάτι τέτοιο. Θα πρέπει να υπάρχει σχετική βούληση και προθυμία. Και αν κάποιος δήμος ή κοινότητα δεν θέλει κάτι τέτοιο, δεν θέλει αυτή τη χειραφέτηση, δεν μπορούμε εμείς να τον αναγκάσουμε, θα χρειαστεί πολύ περισσότερος χρόνος. Τώρα, πώς μπορεί η τοπική διακυβέρνηση να συμβάλλει στην ε, στρατηγική Ευρώπη 2020. Εμείς το κοιτάξαμε υπό τη σκοπιά της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης, αλλά είδαμε και μεμονωμένα παραδείγματα και διαπιστώσαμε ότι υιοθετήθηκαν περισσότερο τέτοιες προσεγγίσεις ε, τοπικής διακυβέρνησης γιατί εστιάστηκαν σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, στις τοπικές και περιφερειακές ανάγκες και είχαν και μία μακροπρόθεσμη προοπτική. Και πολύ συχνά, σε αρκετές περιπτώσεις τουλάχιστον, το τελικό αποτέλεσμα ήταν τελείως διαφορετικό από αυτό, από τις αρχικές προϋποθέσεις. Για παράδειγμα, πολιτικές για την ενεργειακή απόδοση. Πολύ συχνά οι φορείς δεν γνώρισαν καν ότι συνέβαλαν άμεσα στην υλοποίηση της στρατηγικής Ευρώπη 2020. Αλλά το έκαναν, έστω και άθελά τους. Το δικό τους κίνητρο ήταν οι τοπικές αρχές. Είχαν χρησιμοποιήσει, είχαν καθοδηγηθεί από κάποια εγγραφή της ευρωπαϊκό ή της εθνικό ή τοπικό επίπεδο. Αυτό που τους ενδιαφέρει δεν ήταν να συμβάλλουν στην ευρωπαϊκή στρατηγική του 2020, αλλά να συμβάλλουν στην διαμόρφωση της περιφερειακής τους πολιτικής. Αυτά και βάζω τέλεια, για να μπορέσουν και οι συνάδελφοι να πούν κάτι, να πάρουν το λόγο. Σας ευχαριστώ που σταματήσατε, γιατί ούτε δύο λεπτά για τους υπόλοιπους δύο μιλητές δεν περίσσεψαν. Ο κύριος Σούμαν, ένα θέμα θέλω να αναφέρω, μια ερώτηση που επανήλθε πολλές φορές πώς συνδέεται με την Ευρώπη 2020 τοπική αυτοδιοίκηση, γενικότερα πώς συνδέεται ε, με αυτούς τους στόχους. Η απάντηση είναι πολύ σαφή, όσο και σημαντική. Αρκεί να κοιτάξουμε τα μεγάλα μητροπολιτικά κέντρα, τα μεγάλα αστικά κέντρα στην Ευρώπη. Το μισό ΑΕΠ στην Ευρώπη παράγεται στα μεγάλα αστικά κέντρα. Αν δούμε όμως πώς συνδέεται η διακυβέρνηση αυτών των αστικών κέντρων και με τις κοινότητες εκεί, βλέπουμε ότι όταν υπάρχει ένας μεγάλος μετροπολιτικός δήμος που ε, συνδυάζει και συντονίζει τους μικρούς δήμους, είναι πολύ μεγαλύτερη η απόδοση ε, σε σχέση με πόλεις που είναι κατακαιρματισμένες. Και μάλιστα αυτό έχει μετρηθεί κιόλας, 5 με 10% είναι. Τώρα δεν θέλω να μπω ε, σε πάρα πολύ μεγάλες λεπτομέρειες, αλλά αν το έχουμε αυτό υπόψη, το μισό ΑΕΠ μας παράγεται σε πόλεις, ε, μεγάλα αστικά κέντρα, ε, αν το υπολογίσουμε είναι μεγάλα τα νούμερα. Υπάρχει πολύ μεγάλη σχέση λοιπόν με την ανάπτυξη μέσω μακροπρόθεσμα και της πόλης ή την τοπική αυτοδιοίκηση. Και ένα δεύτερο που θα ήθελα να απαντήσω έχει να κάνει με το σωστό επίπεδο αποκέντρωσης ή συγκέντρωσης της διοίκησης. Τι διαπιστώνουμε όταν μελετούμε ε, τις δαπάνες των ε, κυβερνήσεων σε επίπεδο τότερο του κεντρικού. Οι χώρες που το κάνουν αυτό είναι χώρες που έχουν πολύ μεγάλη διοικητική δυνατότητα, με γενικό κρατικό μηχανισμό δηλαδή. Και οι χώρες που υποαπορροφούν είναι χώρες που έχουν αδύναμες διοικήσεις. Και χώρες αυτές δεν έχουν πάρα πολύ καλές επιδόσεις γενικότερα στην οικονομία τους. Θα τους βοηθούσε όμως να μεταφέρουμε μεγάλη ευθύνη σε επίπεδο κάτω του κεντρικού, βεβαίως πάντα ε, στελεχώνοντας αντίστοιχα και ενδυναμώνοντας τη διοικητική μηχανή. Πρέπει λοιπόν να το βλέπουμε έτσι από κάτω προς τα πάνω, να μην κοιτάμε πρώτα τις κυβερνήσεις αλλά το κατώτερο επίπεδο. Αν θέλουμε να αυξήσουμε την αποκέντρωση και να δώσουμε περισσότερες αρμοδιότητες και εξουσίες στις ε, ΟΤΑ, που το θέλει και όσα νομίζω και το υποστηρίζει, αλλά έχει σημασία να αρχίζουμε από το σωστό επίπεδο. Να προσπαθούμε να βελτιώνουμε τη διοικητική τους δυνατότητα και μετά να προχωρούμε. Δεν μπορούμε απλώς να εκχωρούμε αρμοδιότητες, εξουσίες και χρήματα τον προπολογισμό σε κατώτερο του κεντρικού επίπεδου χωρίς να ξέρουμε αν είναι σε θέση να διεκπαιρεώσει αυτές τις αποστολές που του αναθέτουμε. Ευχαριστώ πολύ. Ε, ο κύριος Βαντερλέκ. Για τις περιφέρειες συνέχεια μιλάμε, αλλά δεν έχουμε πάντα χρόνο να δίνουμε το λόγο στις περιφέρειες. Ε, ξέρετε, δεν με πειράζει, τα έχω συνηθίσει αυτά. Ε, τρία σημεία έχω να προσθέσω στις προηγούμενες απαντήσεις των συναδέλφων εδώ. Πρώτον, από τη δική μας πείρα, ε, για το πώς σχεδιάζεις τις διοικητικές δομές και πώς δημιουργείς αρχές. Στη δική μας περίπτωση, κάποια στιγμή καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι και το να ανοίξει κάνει συζήτηση <laughs> δεν θα ήταν δυνατόν. Και πάντα ρωτάμε από ποιον απαρτίζεται αυτή η επικράτεια, σε τι συνίσταται. Δεν είναι μόνο η δημόσια διοίκηση που δεν είναι, αλλά είναι οι πολίτες και οι ιδιώτες επενδυτές. Έτσι χτίζεται μια επικράτεια και αυτό είναι καλό ίσως. Δεν την επιβάλλει μια κρατική οντότητα. Καλό θα ήταν να καταλαβαίνουμε ότι είναι περίπλοκες οι καταστάσεις και δεν μπορούν να ελέγχονται από δομές και κυβερνήσεις μόνο. Διαφωνώ κάπως με το συνάδελφο από τον ΟΣΑ η περιφέρεια δεν είναι κάτι το μονοσήμαντο. Υπάρχουν πολλά πράγματα που επικαλύπτονται και δεν μπορούμε να το ελέγχουμε πάντα από πάνω προς τα κάτω. Εμείς ξεκινήσαμε από κάτω και είδαμε ποιοι είναι οι άνθρωποι που ζουν και δουλεύουν εκεί. Αυτή είναι η περιφέρεια, αυτή είναι η επικράτεια. Να πω και κάτι για τη διοικητική δυνατότητα. Μπορώ από τη δική μου πείρα την προσωπική να πω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό προαπαιτούμενο αυτό. Έχω δει στις δικές μου υπηρεσίες τα 10-15 χρόνια να γίνεται αναδιάρθρωση και αναδιάταξη και βλέπουμε ότι υπάρχουν ικανοί δημόσιοι υπάλληλοι που μπορούν να υπομισθούν ε, αυτό το έργο. Βεβαίως Χρειάζεται κάτι τέτοιο και θα πρέπει να δίνουμε τις ευκαιρίες στους πραγματικούς ανθρώπους που ασχολούνται με αυτά τα πράγματα. Και είναι δύσκολο όταν μιλάμε για κονδύλια και για χρηματοδότηση. Υπάρχουν διαφορετικές κουλτούρες και διαφορετικές νοοτροπίες στις διάφορες δημόσιες διοικήσεις και το θέμα γίνεται πολύ ευαίσθητο και λεπτό. Ένα τελευταίο το οποίο θέλω να αναφέρω είναι αυτή η ιδέα της σημασίας του περιεχομένου. Τι εννοώ Πραγματικά ειλικρινά πιστεύω ότι η ανάπτυξη, ε, η εδαφική και η εδαφική συνοχή έχει σχέση με το περιεχόμενο που της δίνουμε. Και αν υπάρχει κάτι που κάνει την εδαφική συνοχή ή τις εδαφικές πολιτικές πολύ διαφορετικές από τις άλλες, είναι ότι πάντα οι στόχοι είναι κοινωνικοί και είναι πολλαπλοί. Πώς θα συνδέσουμε δηλαδή την κοινωνία και πώς θα βρούμε προστιθέμενη αξία από το σύνδεσμο αυτό. Ακούγοντας τον κύριο Βανίστερ συμφωνώ ότι οι δουλειές, οι θέσεις εργασίας και ανάπτυξη είναι πρωταρχικός στόχος, αλλά από τη σκοπιά της ενταφικής διακυβέρνησης αυτό δεν γίνεται αν δεν το συνδέσεις με τη συζήτηση για την ενεργειακή αποδοτικότητα ή για την κλιματική αλλαγή. Είναι πολλά τα ζητήματα λοιπόν για να υπάρχει ουσιαστική προστιθέμενη αξία και όχι απλώς να δημιουργηθούν κάποιες δουλειές για να έρθει η ανάπτυξη. Αυτή θα είναι μια εδαφική αναπτυξιακή πολιτική. Συνδυάζει πάρα πολλά πράγματα. Πώς να πω, η εδαφική ανάπτυξη δεν είναι από μόνο του ένα ε, στοιχείο, ένα έργο, αλλά η διαχείριση πολλών έργων και ο συνδυασμός τους καταλήγει σε αυτή και την προκαλεί. Εμείς εκεί εστιάζουμε τη χρηματοδότησή μας. Στην προσπάθεια δικτύωσης, συνένωση ανθρώπων, γιατί από αυτούς ζητάς να ξανασκεφτούν, να ξανασχεδιάσουν τις αρχικές τους ιδέες και τα προγράμματα. Αντί να επιλέγουμε λοιπόν ένα έργο να το χρηματοδοτήσουμε, κάπως έτσι λειτουργούμε και θέλουμε να απευθυνθούμε και να απευθυνόμαστε στους ιδιώτες επενδυτές που ξεκινούν από μία ιδέα και το θεωρούν σημαντικό και θεωρούν ότι έτσι παράγεται προς τη θέμενη αξία για την κοινωνία. Σταματώ εδώ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ εκεί Πρόεδρος. Θέλει κανείς να πει τίποτα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Please. Θέλει. Ευχαριστώ. Θα είμαι πολύ σύντομος. Σας ευχαριστώ που μας καλέσατε και θέλαμε να εκφράσουμε την ικανοποίησή μας για την εξαιρετική συνεργασία ε, που έχουμε με την Επιτροπή Ανάπτυξης, ε, Περιφερικής Ανάπτυξης σε σχέση με τις ε, δαφικές προκλήσεις. Πολύ ενδιαφέρουσες οι τρεις σημερινές εισηγήσεις και η συζήτηση που ακολούθησε. Αυτό που θα μπορούσα να προσθέσω είναι ίσως μια διευκρίνηση και κάποια νούμερα που προκύπτουν από τον προγραμματισμό και που ίσως να στηρίξουν τα πορίσματά σας. Από την πρώτη παρουσίαση έγινε μια παρατήρηση που έλεγε ότι η προσημείωση για τη βιώσιμη ανάπτυξη μπορεί να είναι μεγαλύτερη στήριξη για την ευδευτική διακυβέρνηση από τα άλλα μέσα. Θα ήθελα κάπως αυτό να το, ε, να το διευκρινίσω. Το CLD και το ITI είναι ε, μέσα, είναι εργαλεία, ενώ οι ε, είναι συγκεκριμένα ποσά που έχουν αυτή μόνο την κατεύθυνση. Γύρω στο 4% ε, ε, του προϋπολογισμού μπορεί να δαπανηθεί μέσω του ITI και του CLD. Αυτό είναι ένα παράδειγμα ε, λοιπόν και διευκρίνηση για τα νούμερα, αν και οι διαπραγματεύσεις δεν έχουν ολοκληρωθεί με όλα τα κρατημέλη ακόμη. Μάλλον όμως τα νούμερα δεν θα αλλάξουν κατά πολύ το Γενικό Κονδύλι για την Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη έχει ξεπεράσει το 5% που είναι υποχρεωτικό από τον κανονισμό. Φαίνεται να είναι στο 7,58%. Είναι καλύτερο λοιπόν από αυτό που αναμέναμε και για το CLD και το ITI θα πρέπει να, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι είναι προαιρετικά μέσα, δεν επιβάλλονται στα κρατημέλη, ενώ ταυτόχρονα βλέπουμε ότι 17 κρατημέλη χρησιμοποιούν το ITI εκτός της ε, περιφερειακής ανάπτυξης, ε, εκτός συγγνώμη της αστικής ανάπτυξης, οι διάφορες άλλες εδαφικές προκλήσεις, ε, αποτέλεσαν δε αυτά τα δύο μέσα πολύ καλή βάση ώστε να υπάρξει συνεργασία στη χρήση των κονδυλίων. Βλέπουμε πολλά χρήση του ESF και του ERDF. Συνδυάζονται δηλαδή οι, τα διάφορα κονδύλια και οι διάφορες πηγές κονδυλίων. Σας ευχαριστώ πολύ λοιπόν για την προσοχή σας. Σας ευχαριστώ. Οπότε ολοκληρώνουμε τη συζήτηση για το σημείο αυτό. Και το πρώτο σημείο της ημερινής μας ε, μερίσης διάταξης και περνάμε στο δεύτερο θέμα, το Γενικό Προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Δημοσιονομική Χρήση 2016. Όλα τα τμήματα. Η συγκεκριά μας είναι η κυρία Σπυράκη είναι παρούσα. Γνωρίζετε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υιοθέτησε δήλωση προβλέψεων ε, εκτιμήσεων για το 2016 στις 27 Μαΐου και το ενοποιημένο, το σχέδιο προϋπολογισμού στις 24 Ιουνίου και πρότεινε για το κεφάλαιο 1β ε, αναλήψη υποχρεώσεων 51 δις ευρώ και πιστώσεις πληρωμών περίπου 49 δις. 49 δις εκατομμύρια ευρώ. Η Επιτροπή Ρέγγι υιοθετεί κάθε χρόνο γραμμοδότηση για το ψήφισμα που θα συνοδεύει τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ε, τι προτάσει για το προπολογισμό τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Αρμόδια καθήλη για το θέμα αυτό είναι η Επιτροπή προπολογισμών. Σήμερα λοιπόν η συγκεκριά μα, η συντάκτρια τη γνωμοδότησης η κυρία Σπυράκη, θα μα παρουσιάσει το σχέδιο γνωμοδότησης τη. Προτείνω προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών στη γνωμοδότηση την Δευτέρα 27 Ιουλίου του 2015, 5 το απόγευμα. Οπότε, αν εξαρτηθεί αυτή η προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών, μπορούμε να ψηφίσουμε στη συνεδρίασή μας στις 17 Σεπτεμβρίου. Η Επιτροπή Προϋπολογισμών θα ψηφίσει στις 12 με 13 Οκτωβρίου, ώστε αν εμείς ψηφίσουμε νωρίτερα το Σεπτέμβριο, θα μπορεί η γραμματοδοτησή μας να ληφθεί υπόψη από την Επιτροπή Προϋπολογισμών. θα έλεγα να αφιερώσουμε μία ώρα στη συζήτηση για τον προπολογισμό και θα δώσω πρώτα το λόγο στη συντάκτρια της γνωμοδότησης, την κυρία Σπυράκη. Έχουμε τους και ηγητές παρόντες και επίσης και εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από τη Γενική Διεύθυνση Ρέτζιο. Η κυρία Σπυράκη λοιπόν θα είναι η πρώτη μας ομιλητή. Σας ακούμε. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Ε, ασχολήθηκα με την έκθεση λαμβάνοντα υπόψη το σχέδιο προϋπολογισμού για το 2016 και τις ε, συνέπειές του στην περιφερειακή ανάπτυξη. Παρόλο που πρόσφατα έχει οθρηθεί ε, νέος, ε, το νέο σχέδιο προϋπολογισμού, έχουν απομείνει κάποια ζητήματα. Καταρχήν, η στέρηση πληρωμών, οι ανεξόφελτοι λογαριασμοί που θα εμποδίσουν την υλοποίηση κάποιων προγραμμάτων. Διαπίστωσα ότι υπάρχει μείωση του προτινόμενου ποσού σε σχέση με τον προϋπολογισμό του 2015. Αυτό έχει νόημα μόνο σε περίπτωση που το ποσό που προτείνεται θα μπορέσει να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της στέρης πληρώμων και τους ανεξόφλητους λογαριασμού. Για το 2016 όμως έχουμε πιστώσεις ανάλυση υποχρεώσεων που έχουν περάσει από προγράμματα του ε, της προηγούμενης δημοσιονομικής περίοδου και όχι της επόμενης. Ε, οπότε έχουμε αύξηση ε, των πιστώσεων ανάληψη υποχρεώσεων σε σχέση με πέρυσι, αλλά σε ό,τι αφορά την περίοδο 2014-2020 έχουμε κάποιες καθυστερήσεις που κρούν το κόδωνα του κινδύνου σε ό,τι αφορά την, τον κίνδυνο να έχουμε και πάλι ανεξόφλητους λογαριασμούς και συσσόρευσή τους. Μάλιστα, σας παραπέμπω στο σχέδιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που κατά τη γνώμη μου θα πρέπει να δώσει έμφαση στην ενίσχυση της θεσμικής ικανότητας και στη μακροοικονομική εποπτεία. Ευχαριστώ θερμά τους σκιώδης ηγητές και στην εντολή για τον τριμερή διάλογο για τον προϋπολογισμό και περιμένουμε να ανυπομονησία τα σχόλιά σας. Σας ευχαριστούμε κυρία Σπυράκη. Θα δώσω τώρα το λόγο στον κύριο Βόν, που είναι ο σκιώδης ηγετής της ομάδας του. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θέλω και εγώ να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για τις προτάσεις της που είναι σύντομες αλλά σημαντικές και κέρυες. Είμαι ικανοποιημένος που μίλησε για μείωση των πληρωμών στα κατά 4% η Κομισιόν είχε κάνει τη δική της ανάγκηση, ε, ανάλυση και είχε μιλήσει για ένα, ένα για το 1β, 4% μείωση στο 1β είναι παρκές για να ανταποκριθούμε στη ζήτηση του χρόνου. Και αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να το παρακολουθούμε καθώς θα προχωράει η χρονιά. Και βεβαίως η συγκήτρια ανέφερε το ζήτημα των καθυστερημένων πληρωμών το έχουμε συζητήσει επανελειμμένως. Έχουμε καθυστέρηση 20 δις πέρυσι. Η Κομισιόν είπε ότι θα πρέπει να το μειώσουμε με στα 2 δις φέτος. Εγώ δεν ξέρω πώς ακριβώ κατέληξαν σε αυτή τη μείωση, γιατί υπάρχει ζήτηση για τις πληρωμέ και έχω δε επανελειμμένως πει ότι θα ήταν σκόπιμο να ε, δούμε κάποια παραδείγματα προβλημάτων που προκαλούνται λόγω των καθυστερήσεων πληρωμών. Η Κομισογιόν μας έδωσε κάποιες, ε, κάποια παραδείγματα, αλλά και στις περιφέρειες θα πρέπει να υπάρχουν παραδείγματα όπου οργανισμοί και επιχειρήσεις δεν παίρνουν τα χρήματα που χρειάζονται ή, εν πάση περιπτώσει, τα παίρνουν καθυστερημένα λόγω της ε, καθυστέρησης των πληρωμών. Και θα πρέπει αυτά να τα δούμε. Κάτι ακόμα. Έχω και κάτι λεπτομέρειες, αλλά θα τα συζητήσω με την εισηγήτρια. Έχουμε κάνει μεταξύ μας συζήτηση. Ε, Έχω, το θέμα όμως που με απασχολεί είναι αυτό της βασικής χρηματοδότησης, γιατί κάποιες περιφέρειες έχουν προβλήματα για να μπορέσει ε, να προχωρήσουν τα project. Το δεύτερο είναι το νέο ταμείο των στρατηγικών επενδύσεων και πού αυτό μπορεί να παρέμβει. Αυτά λοιπόν και θα ήθελα να συζητήσω και κάποια πράγματα τη με την εισηγήτρια. Άλλοι συνάδελφοι. Κύριε Σκέρλετς. Ευχαριστώ. Αγαπητοί συνάδελφοι, όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, ασχολείται με το θέμα της ε, Ελλάδος και μιλούμε για την ανάπτυξη και τη δημιουργία ε, των θέσεων απασχόλησης. Βέβαια την ανάπτυξη και, ε, και την απασχόληση θα πρέπει να την, τις προωθήσουμε στα πλαίσια της αηφόρου ανάπτυξης. Γι' αυτό και θα πρέπει τα κονδύλια θα πρέπει αυτό το χαρακτηριστικό να έχουν, δηλαδή της αηφόρου ανάπτυξης. Οπότε είναι σημαντικό να μην καθυστερούμε στις πληρωμές, γιατί Πολλά προγράμματα εξαρτώνται από κοινοτικά κονδύλια, οπότε με καθυστερημένε πληρωμέ ή με πληρωμέ απειλείται η υλοποίηση πολλών προγραμμάτων και κυρίω οι μικρομεσαίε επιχειρήσει, οι μικροί τοπικοί δήμοι και κοινότητε, μη κυβερνητικέ οργανώσει είναι οι πιο εκτεθειμένοι και οι πιο ευάλωτοι ε, απέναντι σε τέτοιε καθυστερήσει πληρωμών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να καταβάλουν περισσότερε προσπάθειε και να ενδύνουν την προσπάθειά του για να επιλύσουν τέτοια φλέγοντα προβλήματα, όπω είναι η καθυστέρηση πληρωμών. Ευχαριστώ, κύριο Γιάκοφτσιτ. Σα ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ο κύριο Σκέρλετ και είπε ακριβώ αυτά που ήθελα να πω και μάλιστα στην πανέμορφη κροατική γλώσσα. Δεν πρόκειται λοιπόν να επαναλάβω αυτά που είπε γιατί συμφωνώ μαζί του. Το μόνο που θα μπορούσα να προσθέσω σε αυτά που είπε και η συντάκτρια της γραμματότησης η κυρία Σπυράκη, μία λεπτομέρεια ε, κύριε Βόν και κυρία Σπυράκη. Εμείς ε, ε, δυνάμεθα και γνωρίζω ότι μπορούμε να το κάνουμε και μάλιστα μίλησα και με τον πρόεδρο της Επιτροπής Προπολογισμών, να περιλάβουμε ένα εδάφιο για τη νέα στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι η στρατηγική Αδριατικής Ιωνίου. Συμφωνεί και ο πρόεδρος της Επιτροπής Προπολογισμών. Καλό θα ήταν λοιπόν να ασχοληθούμε με το θέμα αυτό, γιατί και η συγκεκριμένη στρατηγική καλό θα ήταν να έχει κάποια κονδύλια Καλό θα ήταν λοιπόν ακόμη και στην γνωμοδότηση της κυρίας Σπυράκη να πούμε δύο λόγια για την ε, στρατηγική. Αν θέλετε ε, να το βάλετε στην γνωμοδότηση, να δούμε πώς θα εξασφαλίσουμε κάποια κονδύλια που θα χρειαστούν για να εφαρμόσουμε τη στρατηγική για την Αδριατική και το Ιόνιο. Ευχαριστώ. Thank you. Ευχαριστώ. Κυρία Ταμάτο, σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Εγώ ευχαριστώ την ε, συνάδελφο Σπυράκη και συμμερίζομαι την ανησυχία σε σχέση με τη μείωση του 4% των υποχρεώσεων πιστο... Ε, πληρωμών στο 1β. Μιλάμε για πολλά δις λιγότερο από ό,τι σε σχέση με το 14. Δεν ξέρουμε όμως αν θα αρκέσουν για να αντιμετωπίσουμε το σημερινό επίπεδο ε, πληρωμών που προβλέπεται στον τίτλο 1β. Θα πρέπει δεν να καταβληθούν και οι προβλεπόμενες ορισμένες καθυστερήσεις ε, για το, ε, την κατηγορία 1β, δηλαδή 20 δις. Θα πρέπει δεν να αποφύγουμε τα ασφάλματα του παρελθόντος. Γι' αυτό είμαι περίεργη να δω λεπτομερή πρόβλεψη για το πώς θα γίνουν οι πληρωμές ε, στο πλαίσιο της κατηγορίας 1β και επίσης ποιοι είναι οι δείκτες κλειδιά απόδοσης, αν είναι μετρήσιμοι, συγκρίσιμοι και άρα μας λένε κατά πόσο όλα αυτά είναι αποτελεσματικά. Ε, για, το λέω γιατί όπως γνωρίζετε πολύ καλά ένα από τα λάβαρα της νέας πολιτικής συνοχής θα έπρεπε να είναι η δυνατότητα επίτευξης στόχων, συγκεκριμένων στόχων και όχι να δαπανώνται απλά χρήματα και όπου να είναι. Η ίδια η Επίτροπος Κρέτσου μας έδειξε εκείνο το περίφημο χάρτη όπου υπάρχει μια ολόκληρη σειρά περιφερειών όπου εδώ και υπερβολικά πολύ χρόνο δίνονται χρήματα ε, από τα Ευρωπαϊκά Ταμεία αλλά με ισχνά αποτελέσματα. Άρα λοιπόν το θέμα δεν είναι να μειωθούν ε, τα κονδύλια που απευθύνονται σε συγκεκριμένε ε, περιοχέ ή στη στη Συνοχή Ανιγιάννη, αλλά η στη συνοχη εν αλλα η εφαρμογη μια ολόκληρη σειρά δικτών απόδοση που θα μα κάνουν να καταλάβουμε πού έχουμε κάνει λάθο. Και κυρίω να κάνουμε σαφέ για του πολίτε ότι τα αποτελέσματα πρέπει να επιτευχθούν και ότι το πρόβλημα δεν είναι τα χρήματα, αλλά πώ αυτά δαπανώνται. Ε, και κλείνω λέγοντα το εξή. Ε, στη γνωμοδότηση τη συναδέλφου λέει, γίνεται λόγο για την διοικητική ε, ε, ικανότητα. Και μάλιστα είναι κάτι το απαραίτητο στο πλαίσιο τη συζήτησή μα για την περιφερειακή ανάπτυξη. Σα ευχαριστώ. Ο κύριο Έθεριτ έχει το λόγο. Σα ευχαριστώ. Από τότε που μπήκα σε αυτήν εδώ την επιτροπή, Έχω βρεθεί να είμαι κομμάτι αυτής της ταινίας που λέγεται Groundhog Grey. Ε, έχουμε ένα σωρό προγράμματα, ωραία ιδανικά, σχέδια που επηρεάζουν ε, τις, ε, τα διάφορα στρώματα της ζωής, τα διάφορα μάλλον επίπεδα της ζωής, αλλά δεν υπάρχουν χρήματα. Υπάρχουν εκατομμύρια και δισεκατομμύρια, αλλά ποτέ δεν θα αρκούσαν για τέτοιου είδους μεγαλόπνοα και αξιέπαινα προγράμματα. Επαναλαμβάνεται δηλαδή ότι το γεγονός ότι δεν υπάρχουν αρκετά χρήματα για τα σχέδια και τα πλάνα που κάνουμε εγώ πιστεύω πως οι στόχοι είναι πολύ καλοί, αλλά θα πρέπει να γίνονται πολύ συγκεκριμένα πράγματα, κατά τη γνώμη μου, για να βοηθηθούν οι τοπικές οικονομίες. Εάν όμως κανείς θέλει να έχει αυτά τα μεγάλα προγράμματα και να βλέπει αυτά τα τεράστια ποσά, είναι ανεύθυνο όταν ξέρουμε πάρα πολύ καλά από τις συζητήσεις που κάνουμε εδώ πως υπάρχει κίνδυνος για τις εταιρείες που συνεργάζονται ότι να μην πληρωθούν στην ώρα τους. Και ολόκληρο το πρόγραμμα, όσο και φιλόδοξο και αν είναι, μπορεί τελικά να έχει το αντίθετο αποτέλεσμα. Μπορεί τελικά δηλαδή να καταρρεύσουν εταιρείε γιατί δεν πληρώνονται για αυτά που κάνουν. Παρακαλώ λοιπόν θερμά. Ας προσέξουμε λίγο περισσότερο, α φροντίσουμε να μην συμπαρασυρθούμε με όλα αυτά τα υπέροχα που θέλουμε να κάνουμε, α δούμε ποια είναι η πραγματικότητα. Γιατί το πηγάδι με τα χρήματα δεν είναι ανεξάντλητο. Ευχαριστώ, κύριε Σχέτμα. Ευχαριστώ. Και εγώ θα ήθελα να συγχαρώ θερμότατα την ε, κυρία Σπυράκη, που πραγματικά είναι πολύ καλή η έκθεσή της. Θα ήθελα να συγχαρώ θερμότατα την κυρία Σπυράκη για την πολύ καλή της έκθεση. Φυσικά και εγώ με ανησυχία είδα την μείωση ε, κατά 4% των κονδυλίων της πολιτικής συνοχής και Φυσικά ανησυχώ τα μάλα γι' αυτό. Παρ' όλα αυτά όμως θα πρέπει να ακούσουμε τις εξηγήσει της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πώς δικαιολογεί αυτή τη μείωση και πώς θα ξεφύγουμε από αυτό το σπιράλ το, τον της υστέρησης των πληρωμών. Δεν έχουμε χρήματα για να πληρώσουμε ελλημένες υποχρεώσεις. Και τι γίνεται με τι ήδη ενηλυμένε υποχρεώσει που έχουμε από το 2014. Περιμένω με αγωνία τι εξηγήσει Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το σημείο αυτό. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω, θα σας δώσω εντός λίγο το, ρόλο, το λόγο κύριε Βανίσα Ρόι. αλλά ακούγοντας τα σχόλια θα ήθελα να σας υπενθυμίσω την έκτακτη συνεδρίαση της ομάδας εργασίας της Επιτροπής Ρέτζη που επικεντρώθηκε στο πρόβλημα του backlog των πληρωμών, των καθυστερημένων αυτών πληρωμών, των ανεξόφλητων λογαριασμών. Και εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, μας είπαν ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σκοπεύει να αντιμετωπίσει το πρόβλημα αυτό και είμαι γνώμη προς την κυρία Σπυράκη γιατί έλαβε μέρος στην συνάντηση αυτή και είχαμε την ευκαιρία να εξετάσουμε δελεχώς το θέμα και είμαστε έτοιμοι να σας ενημερώσουμε για τις πληροφορίες που λάβαμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη συνεδρίαση αυτή και σίγουρα θα επανέλθουμε στο θέμα αυτό, θα το ξανασυζητήσουμε και είμαστε έτοιμοι να οργανώσουμε και νέα τέτοια έκτακτη συνεδρίαση με πιο ευρία συμμετοχή των μελών της Επιτροπής. Πάντως θα σας στείλουμε τις πληροφορίες ε, που ετοιμάστηκαν από τις υπηρεσίες Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ειδικά για τη δική μας Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης. Αυτά και να δώσω το λόγο στον κύριο Μπρούα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Το σχέδιο γνωμοδότησης μιλάει για μείωση των πιστώσεων πληρωμών στο 1β για την ανάπτυξη και στις πιστώσεις πληρωμών στο προσχέδιο προϋπολογισμού του 2016 είναι συγκρατημένη αύξηση 1,06%. Ε, Το θέμα της ευφυούς ανάπτυξης και περνάει από 51 δις σε 49, δηλαδή έχουμε μια ε, μείωση 4% ουσιαστικά. Αυτή η μείωση θα έρθει να επιδεινώσει ε, τους ανεξόφλητους λογαριασμούς που έχουν ε, φτάσει σε σημείο ρεκόρ. Αυτό μας ανησυχεί διότι και όλοι το γνωρίζουν εδώ διακυβεύονται στα κράτη-μέλη οι οργανισμοί διαχείρισης των επιχειρησιακών προγραμμάτων και επίσης οι φορείς που ενέχονται κινδυνεύουν από τις καθυστερημένες πληρωμές. Κινδυνεύει επίσης η Ευρωπαϊκή Ένωση να χάσει την αξιοπιστία της, γιατί πρόκειται για την αναδιανομή δημοσίου χρήματος ε, που εμφανίζει τις λειτουργίες και βλέπουμε ότι υπονομεύονται και τα σχέδια σε τοπικό επίπεδο είναι πάρα πολύ απαραίτητα για τους πολίτες. Πώς θεωρείτε λοιπόν ότι οι περιφέρειες θα καταφέρουν να αντιμετωπίσουν αυτή την υπερημερία στις πληρωμές αυτό προφανώς θα επηρεάσει και τις άλλες θέσεις του προϋπολογισμού που έχουν σχέση με τις αρμοδιότητες των περιφέρειων. Ενώ όλοι στην Ολομέλεια χαίρονται και ε, χειροκροτούν την δημιουργία θέσεων εργασίας από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, εδώ δυστυχώς κανείς δεν θορυβείται από ε, την κατάσταση αυτή γιατί χρειάζονται χρήματα μικρομεσαίες για να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας. Και αυτό που είναι το πλέον απίστευτο είναι ενώ στο σχέδιο προϋπολογισμού γενικά βλέπουμε μείωση για το 2016 των πιστώσεων πληρωμών υπάρχουν άλλες θέσεις του προϋπολογισμού όπου τα κονδύλια τους αυξάνουν ε, εντυπωσιακά στην πρικοδότηση. Και εδώ εννοώ την ασφάλεια και τους ε, πολίτες ε, που έχει αύξηση κατά 17% για να αντιμετωπίσουμε υποτίθεται ε, ε, τη ροή παράνομων μεταναστών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και επίσης αυξάνεται και η χρηματοδότηση της εξωτερικής πολιτικής Ένωσης κατά 28% παρακαλώ φέτος ή οι διοικητικές δαπάνες που αυξάνονται επίσης κατά 20%. Αυτές είναι κάποιες ανησυχίες που θα ήθελα να μοιραστώ μαζί ε, σας στην Επιτροπή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Τώρα και ο Σβανίστε Ρόη. Πρόεδρε, ε, Σύμφωνο με τις ε, παρατηρήσεις που έγιναν γενικότερα. Ενδεχομένω το σημείο 1 θα μπορούσε να έχει οξύτερη διατύπωση, ε, εκτός από την ανησυχία, ίσως να μιλήσουμε και για κατάσταση που μας έχει θορυβήσει, όχι απλώς ανησυχήσει και μπορούμε να το συνδέσουμε αυτό το σημείο με το δεύτερο άρθρο γιατί όταν ε, είναι συνεχώς λιγότερα τα χρήματα, δεν βγαίνει ο λογαριασμός από μηχανής, δηλαδή πώς θα έρθει η λύση. Και τα κράτη-μέλη, ε, ορισμένα από αυτά, εν πάση περιπτώσει, δεν μπορούν να υλοποιούν τα προγράμματά τους. Ε, κάτι πρέπει να γίνει όταν κόβονται τα κονδύλια σε αυτό το πρόγραμμα δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ε, πρέπει να δούμε ε, με τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό τι γίνεται με τα οικονομικά μας και πώς αυτά πληρώνονται. Πώς θα λυθεί το πρόβλημα. Το 2015 δεν υπήρξε καμία βελτίωση. Τέλη του 2015 έχουμε περίπου 20 δισεκατομμύρια. Και τι θα γίνει επαναστατικό για να μειωθεί το νέο πρόγραμμα συνεχίζει και προχωράει, αλλά ε, θα πρέπει να είμαστε περισσότερο από ανήσυχοι. Ε, θα πρέπει να πούμε ότι αγωνιούμε, βάση περιπτώσει, γιατί κινδυνεύουν τα προγράμματα. Και ένα δεύτερο, θα μπορούσε η Πρόεδρος να μας πει πόσο έχει προχωρήσει η Επιτροπή Οικονομικών με το πρόγραμμα αυτό Καλό είναι να κάνουμε εμείς νομοδοτήσεις, το έχουν συνηθίσει αυτοί, αλλά δεν είναι ε, ικανοποιητικά τα όσα συνέβησαν το 2015. Υπάρχει το επιχειρησιακό πρόγραμμα και θέλω να ε, συμμετέχουμε και εμείς βεβαίως, αλλά να πούμε ότι ανησυχούμε βαθύτατα και να δούμε ποιες είναι οι επιπτώσεις. Αν δεν καταφέρουν τα κράτη-μέλη να αντισταθμίσουν αυτές τις καθυστερήσεις με την επικουρικότητα κτλ. Θα είναι πολύ αρνητικά όλα τα αποτελέσματα. Γενικά θαυμάζω την κυρία Σπυράκη που κάθεται εδώ με τέτοια ηρεμία και δεν ε, είναι ε, ε, η σκέψη της και το μυαλό της αλλού. Όταν μπήκα τη ρώτησα αν, κοιμήθηκα, αν κοιμήθηκε τη νύχτα και μου λέει όχι δεν κοιμήθηκα, μάτι δεν έκλεισε με όλα αυτά που συμβαίνουν στην Ελλάδα. Ευχαριστώ πολύ. Thank you. Thank you very much. Σας ευχαριστώ. Άλλος κανείς. Όχι, οπότε θα δώσω το λόγο στον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ο κύριος Τουμπελουίτσκι, ή κάπως έτσι. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να σταθώ σε δύο σημεία. Το ένα είναι αυτό που αναφέρατε ήδη και εσείς. Είχαμε την ε, ομάδα εργασίας για το θέμα του σχεδίου χρηματοδότησης ε, για να καλυφθεί το θέμα των καθυστερημένων των υπερημένων πληρωμών. Και έχει ήδη προταθεί το σχέδιο προπολογισμού προκειμένου να αντιμετωπιστούν καθυστερημένε πληρωμέ ε, για την περίοδο 2014-2020. Πιστεύουμε ότι θα ε, λύσουμε το πρόβλημα της προηγούμενης περίοδου 2007-2013 και το 2016 αρκεί να μην γίνουν περαιτέρω περικοπές στον προϋπολογισμό. Και δεδομένων των προβλέψεων πληρωμών ε, για την περίοδο 2014-2020 από τα κράτη-μέλη θα τηρηθεί. Και στην προηγούμενη περίοδο έληξαν κάποια προγράμματα και γι' αυτό έχουν ε, μείνει ανεξόφλητοι κάποια, κάποιοι λογαριασμοί που πέρασαν σε, στην επόμενη περίοδο. Πιστεύουμε ότι το σχέδιο προπολογισμού προβλέπει αρκετέ πιστώσει πληρωμών για να απορροφηθούν οι καθυστερημένε πληρωμέ και να πληρωθούν οι ανεξόφλητοι λογαριασμοί μέχρι το τέλη του έτου και την επόμενη χρονιά. Τώρα, για τις πληρωμές, για τις καθυστερημένες πληρωμές. Προς το παρόν μπορώ να σας ε, διαβεβαιώσω ότι μέσα 16 μέρες ε, πληρώνονται οι αιτήσει που υποβάλλουν το κράτη-μέλη από τη Γενική Διεύθυνση Ρέγγιο και μετά τις διαπραγματεύσει ε, για την επόμενη περίοδο προγραμματισμού 2014-2020 κάνουμε ό,τι μπορούμε για να αποφύγουμε στο μέλλον τέτοια συσσόρευση ανεξόφλητων λογαριασμών αλλά υπάρχουν, υπάρχει το σύστημα των διαφορετικών φάσεων ε, πληρωμών που ισχύει και για την επόμενη περίοδο με τακτική ροή εκεί. και θέλουμε φυσικά να εξασφαλίσουμε ε, κονδύλια συνεχώς για τους δικαιούχους των προγραμμάτων για να μην ε, χρειαστεί να σταματήσουν τα προγράμματα. Παρακολουθούμε λοιπόν εκ του σύνεγγυς τις διαπραγματεύσεις για τον προϋπολογισμό του επόμενου έτους. Σας ευχαριστώ. Κύριε Σπυράκη. Εσείς τώρα θέλετε να δευτερολογήσετε, θέλετε να απαντήσετε. Όπως σας είπα πρόεδρε, θα περιμένω τις τροπολογίες των συναδέλφων και φυσικά θα λάβω υπόψη τα όλα όσα υπόθηκαν εδώ. Ευχαριστώ. εγώ σας ευχαριστώ όλους όσοι συμμετείχατε στη συζήτηση. Να σας θυμίσω ότι 27 Ιουλίου στις 5.30 το απόγευμα είναι η προθεσμία επιβολής τροπολογιών για το σχέδιο αυτό γνωμοδότησης και θα ψηφίσουμε στις 17 Σεπτεμβρίου για την τελική εκδοχή της νομοδότησης. Τώρα, συνεχίζουμε με την ημερήσια διαμεδιάταξη. Έχουμε συνεδρίαση των συντονιστών. Οι υπόλοιποι συνάδελφοι θα τα πούμε αύριο το πρωί στις 9.